So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und recht herzlich willkommen zu unserer Κυρίες και κύριοι, ε, σας καλωσορίζουμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 1 της σημερινής διάταξης, την οποία και θα εγκρίνουμε με δύο τροποποίησεις. Ε, είναι το σημείο υπαριθμών 6 και το υπαριθμών 7. Αυτά αναβάλλονται αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα άλλο στην ημερήσια διάταξη που σήμερα είναι πολύ φορτωμένη. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει να είμαστε ε, αρκετά ε, σύντομοι στις παρεμβάσεις μας ε, οι συγητές και οι συνεισηγητές αν δεν τα αν δεν τηρήσουν το χρόνο, δεν θα μπορέσουν ε, να λάβουν όλο το λόγο. Και όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες, νομίζω ότι έχουμε ανακοινώσει το πόσο χρόνο έχουν. Θα τους το ξαναεπενθυμίζω. Έχουμε σήμερα όλες τις γλώσσες, εκτός από φινλανδικά, μαλτέζικα, κροατικά και ε, γκέλις. Ο Ντέιβιτ δεν είναι σήμερα παρόν, αλλά βεβαίως και θα λάβω υπόψη ότι όλοι εσείς διαμαρτύρεστε. Εγκρίνουμε λοιπόν τα πρακτικά ε, της 18ης, 19ης ε, Απριλίου, 12 Ιουλίου και 13-14 Ιουλίου. Ε, προσθήκες δεν υπήρξαν επ' αυτού, ούτε και αλλαγές. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 4 της ημερήσιας διάταξης. Σε αυτό το σημείο Ήδη στα γερμανικά ο τίτλο είναι πάρα πολύ περίπλοκος. Προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσει προσβασιμότητα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ε, τα έχετε αυτά στα αγγλικά ε, μπροστά σας. Σήμερα έχουμε και μία ακρόαση για 45 περίπου λεπτά και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τους εμπειρογνώμονες που έχουμε προσκαλέσει. Με τους εμπειρογνώμονες θέλουμε να συζητήσουμε και ε, στην ε, περίπτωση αυτή ας μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και, υπάρχουν και οι διαφάνειες που θα προβάλλονται που διευκολύνει. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω θερμά τους ε, εμπειρογνώμονες Ingrid Heindorf ε, που είναι συντονίστρια στη Γενέβη, τον κύριο Ντέβιτ Καπότσι, ο οποίος είναι εκτελεστικός ε, διευθυντής, Σαμπίνε Λούμπνικ, Mobile Manufacturers Forum, και επίσης ε, να καλωσορίσω και την κυρία Άννα Λόρσεν που έρχεται από το Πανεπιστήμιο του Λίτς, ε, καθηγήτρια ε, νομικής. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους θερμά. Και χωρίς τις τίποτα παραπάνω, χωρίς να προσθέσουμε τίποτα παραπάνω, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τις ε, παρουσιάσεις. Ε, σήμερα, όπως σας είπα, είναι πολύ φορτωμένη η μερίσια διάταξη, γι' αυτό λοιπόν, αν τηρείτε τα 7 λεπτά, θα σας είμαι ευγνώμων. Η κυρία Ingrid Χάιντορφ είναι η πρώτη εμπειρογνώμων και της δίνω και το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που μας προσκάλεσαν να συμμετέχουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό event. Είμαστε μια οργάνωση πολύ σημαντική για άτομα με αναπηρία. Έχουμε τρεις στόχους να παρακολουθήσουμε την κατάσταση του CRPD, για την αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, και προσπαθούμε να προωθήσουμε γενικές λύσεις, βασιζόμαστε στην προσβασιμότητα, στη συμμετοχή στα πολιτικά δρόμενα, εκπαίδευση, τεχνολογίες των πληροφοριών και άλλα. Οι προσβάσιμε τεχνολογίε και υπηρεσίε είναι προπόθεση για να μπορεί κανείς να απολαμβάνει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προσβασιμότητα είναι ζήτημα σε και θανάτου. Το 2014 η μα έδειξε ότι στι περισσότερε χώρε που ερευνήσαμε δεν υπήρχαν ε, επαρκή συστήματα έγκαιρης προειδοποίηση ε, προσβάσιμα ή γραμμές ε, τηλεφωνικές προσβάσιμες. Από το 2011 βλέπουμε στη, με, τον σεισμό στην Ιαπωνία ότι αν υπήρχαν αυτές τις τεχνολογίες θα μπορούσαν να χάσουν πολλά άτομα με αναπηρία το έχασαν τη ζωή τους. Η UNESCO τώρα θεωρεί ότι πρόσβαση στη γνώση ε, με τη βοήθεια των ε, αποβρεθόμενων από τεχνολογία από την πληροφορική τεχνολογία είναι ένα αναπαρατήριο το ανθρώπινο δικαίωμα. Έχουμε το ίντερνετ, τα κομπιούτερ, τα smartphone, ε, τις ταπλήτες. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ιντερνετικά μαθήματα για τις προσβάσιμες τεχνολογίες. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά σας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. <laughs> <laughs> Ναι, είμαι έτσι λίγο... Με έχει συνεπάρει ο ενθουσιασμός, βλέπετε. Έτσι λοιπόν οι προσβάσιμες τεχνολογίες βελτιώνουν μεταξύ άλλων και την απασχολησιμότητα. Μπορεί ο κόσμος να εργαστεί το 2013 η ερευνά μας έδειξε ότι έλλειψη προσβασιμότητας στο χώρο εργασίας, στις εκπαιδευτικές ε, καταστάσεις, στις ε, συγκοινωνίες είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους θα πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις ε, δομές που μέχρι στιγμής δεν είναι επαρκείς. Αλλάζουν τα πράγματα, όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται ψηφιακή τεχνολογία. Με βάση τον ΩΣΑ, το 25% ε, των θέσεων εργασία αλλάζουν λόγω τη αυτοματοποίηση. Η προσβασιμότητα είναι για όλου ε, και είναι και ευκαιρία και για του οικονομικού φορεί. Θεωρείται όμω ακόμη ω αποκλειστικό όφελο για τα άτομα με αναπηρία. Δεν ισχύει αυτό. Η προσβασιμότητα ωφελεί όλα τα μέλη τη κοινωνία. Η μη προσβασιμότητα αφορά τα παιδιά, τις εγγύους, τους τουρίστες, τους μετανάστες, τους ηλικιωμένου. Μεταξύ του 2015 και 2014 με τη Βιεντέζα, οι άνω των 60 ετών θα έχουν αυξηθεί κατά 5%. Κατά 56%. Βλέπουμε ότι με την προσβασιμότητα θα μπορούσαν να υπάρξουν και οικονομικά ωφέλη. Κρατήσεις, ηλεκτρονικές, ε, πιο σαφή τα μενού, λιγότερες καταγγελίες ε, κτλ. Κάποια βασικά μηνύματα λοιπόν, τα οποία προέκυψαν από την έρευνα τώρα, ένα νομικά δεσμευτικό μέσο συνιστά πλεονέκτημα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πλήρης διάσταση και του κόστους του, της προσβασιμότητας η κοινωνική, συμπεριφοριστική επικοινωνία, η, αξι... η φυσική οικονομική προσβασιμότητα έχουν προβληθεί με το Zero Project, ε, για παράδειγμα, τονίσαμε και την νοητική διάσταση που πολύ συχνά παραγνωρίζεται. skills and those 75 million European adults who have low qualifications Θα βοηθηθούν οι άνθρωποι λοιπόν με τις νοητικές ε, ανεπάρκειες και αδυναμίες ή και πολλά παιδιά, ένα στα πέντε κάτω των 15 ετών που έχουν προβλήματα. Όλες οι υπηρεσίες και τα πέντε θα πρέπει να είναι προσβάσιμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν όλοι στο μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς να χρειάζεται μεγαλύτερη προσαρμογή να υπάρχουν κάποια εξειδικευμένα χαρακτηριστικά. Θέλω να σας ε, συγχαρώ όλους όσους έχετε συνεισφέρει στο σχέδιο αυτής της δράσης για την προσβασιμότητα. Και στηρίζω και αυτό το φιλόδοξο πλαίσιο για την προσβασιμότητα σε σχέση με προϊόντα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Nun darf ich das Wort geben Herrn David Capozzi vom US Access Board. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Καπότσι παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να έρθω εδώ. Έχω πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα της αναπηρίας. Ήμουν ένας από τους εννέα νομικούς ε, που ε, συμμετείχε σε μια εξειδικευμένη ομάδα ακριβώς για αυτό το νομοσχέδιο περί αναπηρίας ε, που έχει ε, καταθέσει πάνω από 20 νομοσχέδια, νομικές προτάσεις ε, για το θέμα της ε, αναπηρίας και καλύπτουμε και ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Και έτσι με αυτή την εμπειρία παρέχω τα σχόλιά μου για, τα, για τέσσερις τομείς σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό πακέτο ε, εδώ της προσβασιμότητας και τα δικά μου σχόλια και τη δική μου κυβέρνησης. Πρώτον, σα συγχαίρουμε γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το θέμα της προσβασιμότητα ε, σε ορισμένα εμπορεύματα και υπηρεσίε. Παρ' όλα αυτά, με εκπλήσει το περιορισμένο πεδίο εφαρμογή ε, του νομοσχεδίου. Ε, συνήθως μιλούμε μόνο για την δημόσια πρόσβαση, μέσα μεταφοράς, κτίρια, υποδομές κτλ. Ε, ο δικός μας φορέας έχει προϋποθέσεις ε, υποδομών ε, ευρύτερα και για τα κτίρια, τα ομοσπονδιακά, κρατικά και ιδιωτικά τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτό περιλαμβάνουμε από τα δικαστήρια, τα εστιατόρια, θέατρα, γραφεία, παιδικές χαρές, πισίνες, αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκα αναψυχής, πάρκα και παραλίες. Και τώρα οριστικοποιούμε νέε προποθέσει για τα μονοπάτια, τις ράμπες, τις διαβάσεις, ε, τα πάρκινγκ μαζί και με νέε προποθέσει για τις διαγνωστικές, ε, διαγνωστικό εξοπλισμό. Και η πρόταση νόμου, όταν δεν συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα, είναι ελλειπής. Δεύτερον, ε, τίθενται όλε αυτές οι προποθέσει σε λειτουργικό επίπεδο. Δεν έχει πάει τόσο καλά αυτή η προσέγγιση στις ΗΠΑ. Το 1991 είχαμε τις κατευθυντήρες γραμμές ε, για τους Αμερικανούς με αναπηρία και εκεί είχαμε συγκεκριμένες ε, αυτοματοποιημένες ε, μηχανές, εξοπλισμό και ανέφερε ότι οι οδηγίες και όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να δίδονται, να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση και σε άτομα με περιορισμό στην όραση. Όμω αυτό ήταν τόσο ασαφές που τελικά είχαμε κάποια ATMs με οδηγίε Braille πάνω στι ε, πλάκε αυτέ, αλλά χωρί καμία αλλαγή στο λειτουργικό σύστημα των ATM. Και έτσι δεν μπορούσαν ε, ε, οι τυφλοί να τα χρησιμοποιήσουν. Επομένω, οι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των τυφλών πραγματικά αγανάκτησαν και απέτησαν να υπάρχει και ακουστικό υλικό. Στη συνέχεια το δικαστήριο απεφάνθη ότι ήταν τόσο ασαφείς οι οδηγίες μας ε, και ότι έτσι δεν, δεν ήταν απαραίτητο το, οπτικό, το ακουστικό συνομή υλικό και γι' αυτό το 2004 ε, αναθεωρήσαμε τις καθημερινές γραμμές για να παρέχεται και ακουστικό υλικό από τα ATM. Έχουν συγκεκριμένο ε, σχεδιασμό στο πληκτρολόγιο και έχουν και υποδοχή για ακουστικά. Πάνω από 100.000 τέτοια ATMs έχουμε πλέον στις ΗΠΑ. Τα πρότυπά σε ό,τι αφορά την ε, τεχνολογία της πληροφορίας περιλαμβάνει περίπου αυτά που αναφέρετε κι εσείς και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα ε, πρότυπα λειτουργικών επιδόσεων. Όμω, απαιτούμε και μετρήσιμα τεχνικά πρότυπα και τα δύο. Αν υπάρχουν τεχνικέ διατάξει που αφορούν ένα προϊόν, τότε δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανεί τα κριτήρια λειτουργική επίδοση. Αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για την γενική αξιολόγηση ποιότητα ε, του ε, προϊόντος και για τεχνολογίε όπου δεν υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα. Μόνο όταν ένα προϊόν δεν καλύπτεται πλήρω από τι τεχνικέ διατάξει, τότε εξετάζουμε τα κριτήρια λειτουργική επίδοση. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιούμε τα πρότυπά μα ICT και τα εναρμονίζουμε με τα νέα πρότυπα ε, EN301 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει και τα ε, κριτήρια λειτουργικών επιδόσεων και τα τεχνικά κριτήρια, όπως και τα δικά μας πρότυπα. Σε συνδυασμό και με, με το παράρτημα 1 και πάλι θεωρούμε ότι καλύτερο θα ήταν να χρησιμοποιηθεί το EN ως ε, σημείο αφετηρία στην προσβασιμότητα και καλό θα ήταν να ενισχυθεί και αυτό το EN. Τρίτον, καλό θα ήταν να είστε προσεκτικοί σε τη φορά τη χρήση σήματος για την ε, αναφορά προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και εμπορεύματα Ιδίω όταν τίθενται προποθέσει μόνο σε λειτουργικό επίπεδο. Γιατί είναι δύσκολο να μετρήσει κανεί ε, αυτέ τι λειτουργικέ προποθέσει, όπω είναι το παράδειγμα του ATM. Αυτό που ένα κατασκευαστή θεωρεί ε, προσβάσιμο, δεν το θεωρεί ε, προσβάσιμο ένα άλλο. Σε συνδυασμό με το σήμα CE, μπορεί να είναι και παραπλανητικό για του καταναλωτέ. Τα ATM, για παράδειγμα, θα πρέπει να δίνουν τρόπου λειτουργίε με ε, Συγκεκριμένε προϋποθέσεις. Ε, για παράδειγμα τα 12 εκατοστά από το έδαφος. Όμως αυτό είναι αυθαίρετο. Ποιος κρίνει ποιο είναι το κατάλληλο ύψος ή βάρο ε, και ούτω καθεξής. Οι κατασκευαστές λοιπόν μπορούν να, να επιλέξουν οποιαδήποτε δυνατότητα και να θέσουν το σήμα. Εμείς δεν απαιτούμε σήμα για τα προϊόντα ICT υπό το δικό μας νόμο ακριβώς για αυτό το λόγο. Και τέλος, ε, σας παροτρύνω να έχετε ένα εύρωστο σχήμα επιβολής του νόμου γιατί απαιτείται σημαντική προσπάθεια. Η δικοί μα νόμοι προσβασιμότητα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στι ε, πολιτικέ μα ελευθερίε και τέτοιε αρχέ, ε, σε παράπονα, αστικέ κυρώσει ε, και το Καλό είναι λοιπόν να τα παίρνουμε και με τη σειρά τα πράγματα, όμω αν δεν έχετε έναν συνολικό εύρο στο μηχανισμό επιβολή του νόμου, κατά πάσα πιθανότητα θα, ε, θα αποτύχει το νομοσχέδιο και όλη η προσπάθεια. Πρέπει να υπάρχουν ένδεκα μέσα, αλλιώ δεν προστατεύονται τα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Σαμπίνε ε, Mobile Factors ε, Forum. Εγώ έχω, προετοιμάσει μία ε, ομιλία με PowerPoint. Yes, perfect. Many thanks. First of all, a big thank you for inviting us here to share. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλείτε για να ακούσουμε τα σχόλιά σας ε, για αυτό το, την πράξη προσβασιμότητας. Εγώ εκπροσωπώ μια Ένωση που ασχολείται με τον σχετικό εξοπλισμό και έχουμε δουλέψει για την κινητή προσβασιμότητα για πάνω από 8 χρόνια και τα αποτελέσματα ε, ήταν να προκύψει μια ε, τράπεζα δεδομένων ε, η οποία δίνει δυνατότητα για πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνο, σε τάμπλετ και σε άλλα παρεμφερή, άλλες Σήμερα Έχουμε περίπου 1.200 κινητά με αυτά τα στοιχεία της προσβασιμότητας ε, και σε πάρα πολλές ε, γλώσσες. Τώρα, όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθετική Πράξη Προσβασιμότητας, θα ξεκινήσω με ένα θετικό μήνυμα ότι στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να προάγει την προσβασιμότητα και να βελτιώσει περαιτέρω την προσβασιμότητα. 18 εταιρείε που ε, εμπλέκονται σε αυτό το πρόγραμμα έχουν ε, δεσμευτεί να ε, βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σήμερα και επίσης να έχουν και μία άμεση ανταλλαγή απόψεων με τους χρήστες. Βασικός στόχος του προγράμματος Gary είναι να βελτιωθούν οι πληροφορίες για ήδη υπάρχουσες λύσεις, καλύτερες πληροφορίες προς τους καταναλωτές και να τους δώσουν τη δυνατότητα να βρουν τη συσκευή που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους. Και βεβαίως αν υπάρχουν ε, τα στοιχεία αυτά της προσβασιμότητας το ένα δίπλα στο άλλο, αυτό προφανώς και βελτιώνει και τον ανταγωνισμό. Ε, θα ήθελα τώρα να αφαιρθώ σε δύο στοιχεία, τα οποία ανέφερε ήδη ο Ντέιβιτ στην ομιλία του, ε, ο e και η functional approach. Όσον αφορά το ε, λογότυπο CE, νομίζω ότι εάν πρόκειται να χρησιμοποιείται για θέματα προσβασιμότητας, πολλοί κατασκευαστές θα μπορούσαν να πούνε ναι, πράγματι ε, αυτό η συσκευή είναι προσβάσιμη και μπορώ να τοποθετήσω το λογότυπο ή όχι. Αλλά η προσβασιμότητα δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω δύο πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα για να σα εξηγήσω τι ακριβώ εννοούμε. Έχουμε λοιπόν ε, στην ε, οθόνη δύο συσκευέ τη συσκευή A που έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά που την καθιστούν προσβάσιμη για άτομα με περιορισμένη ορατότητα. Ε, μεγενθύνεται η ε, οθόνη, πάρα πολλά ε, χαρακτηριστικά. Όμως ε, δεν έχει έναν προεγκατεστημένο screen reader ε, και έτσι αυτό η συσκευή δεν είναι προσβάσιμη για άτομα χωρίς καθόλου όραση. Η συσκευή Β όμως είναι προσβάσιμη για άτομα με περιορισμένη ακοή, έχει ε, την συμβασιμότητα με text phone, αλλά εκείνο που δεν έχει είναι δεν έχει βελτιωμένη ποιότητα των ακουστικών. Άρα ε, δεν είναι προσβάσιμη για αυτούς που δεν έχουν σχεδόν καθόλου ακοή. Και με βάση την προσβασιμότητα και τη σχετική νομοθετική πράξη, καμία από αυτές τις δύο συσκευές δεν μπορούν να απολυθούν στην αγορά, γιατί το το, ο λογότυπος είναι απόλυτος όταν χρησιμοποιείται. Παρότι λοιπόν αυτές οι συσκευέ ε, ε, είναι κατά κάποιο τρόπο προσβάσιμες, δεν μπορούν να τεθούν στην αγορά. Τώρα, όσον αφορά τη λειτουργική προσέγγιση, εμείς ε, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί με την έννοια ότι στο παράρτημα 1 ε, πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές για εναλλακτικά χρώματα. Η λειτουργική προσέγγιση, όπως αναφέρεται και στις ε, προδιαγραφές 3.01.549 που ανέφερε και ο Ντέιβιτ, ε, εκεί προβλέπεται ότι τουλάχιστον ένα στοιχείο, η μία συσκευή δεν θα απαιτεί χρώμα από το χρήστη, να μπορεί να κατανοεί, να βλέπει το χρώμα. Ε, θέλω λοιπόν να σας πω ότι εμείς έχουμε τον κοινό στόχο του να δίνουμε δυνατότητα χρήστης, χρήσης στο χρήστη, αλλά και ο κατασκευαστής να ενημερώνει τον καταναλωτή, να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τις λύσεις που μπορούν να υπάρξουν στην αγορά σήμερα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια λειτουργική προσέγγιση και εμεί σας συστήνουμε να ε, επικεντρώσουμε την προσοχή μας περισσότερο στις αναφορές ε, στις εκθέσεις και όχι τόσο στο λογότυπο. Για λόγους χρόνου ε, δεν μπορώ να αναφερθώ σε περισσότερα στοιχεία, αλλά υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι το να χρησιμοποιούμε αυτό το λογότυπο δεν μας βοηθά. Και τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι ε, είμαστε πολύ ευτυχείς ε, που συνεργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο για να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο και μάλιστα να βρούμε τον τρόπο να τον επιδιώξουμε από κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, Άννα Λάρσεν από το Πανεπιστήμιο Leeds, παρακαλώ. Okay, many thanks, Chair, and... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει ένα πολύ περήφανο μικρό ιστορικό για την πρόθεση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία. Σήμερα θα σας μιλήσω για τις ε, νομικές ε, ανάγκες και ε, ευκαιρίες και το ηθικό ζήτημα που άπτεται αυτής τη Ευρωπαϊκή νομοθετικής πράξη για την προσβασιμότητα. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι, ποιες είναι οι νομικές απαιτήσεις. Έχουμε τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία. Σε απειντή. Έχει επικυρωθεί, όπως γνωρίζετε φαντάζομαι, από την ευρύτατη πλειοψηφία των κρατών μελών. Μόνο ένα δεν την έχει ακόμη. Όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά δεν την έχει ακόμη υπογράψει. σε ό,τι αφορά το αρμογή των υποχρέωσεων της RPD, ε, υπάρχει επιτροπή παρακολούθησης του ΟΗΕ που είδε ε, το τι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και αναγνωρίζει τη σημασία της ε, νομοθετική πράξης για την προσβασιμότητα που καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να την εγκρίνει το στομότερο δυνατό. Κύριο στο άρθρο 9 της συνθήκης CRPD θεσπίζονται αυτές οι υποχρεώσεις. Τα συμβαλόμενα μέρη λοιπόν θα πρέπει να δίνουν ισότιμη πρόσβαση για μεταφορές ε, στους, στις διάφορες υποδομές, πληροφορίες, επικοινωνίες και τεχνολογίες πληροφοριών, επικοινωνιών και συστήματα και οτιδήποτε άλλο διατίθεται στο ευρύ κοινό. Τόσο στην Ήπεθρο και στις αστικές περιοχές θα πρέπει να εντοπιστούν και να παλιφούν τα εμπόδια, οι φραγμοί, να υιοθετηθούν ελάχιστα πρότυπα, κατευθυντήρες γραμμές και να προωθηθεί ο σχεδιασμός, όπως επίσης και να προωθούν οι προσβάσιμες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Αυτό είναι το άρθρο 9. Και σε άλλα άρθρα αναφέρονται σχετικά με την προσβασιμότητα. Ε, ζητήματα είναι όμως και μια από τις βασικές αρχές που διατρέχει όλη την σύμβαση, CRPD. Δηλαδή πρόκειται για ένα εγκάρσιο ζήτημα Είναι δικαίωμα η προσβασιμότητα. Γιατί αλλιώ χάνουν το νόημά του για πολλού ανθρώπου με αναπηρία τα ανθρώπινα δικαιώματα συνολικά. Κάτι τελευταίο για την σύμβαση, για το CRPD, είναι το άρθρο 4.3. Εκεί ζητείται η διαβούλευση με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία για την υλοποίηση πολιτικών που αποσκοπούν στην εφαρμογή της σύμβασης. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα πλαίσια. Τώρα περνάμε στις νομικές ευκαιρίες. Έχουμε λοιπόν αυτή την επιτακτική ανάγκη αφενός δεσμεύσει ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως και οι Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να τα προωθούν. Τώρα, μέσω τη Ευρωπαϊκή Νομοθετική πράξη για την προσβασιμότητα δίνεται δυνατότητα, τη ευκαιρία να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερική αγοράς. Ούτε να δημιουργηθούν οι θεσμοί, αλλά και να απαλληφθούν οι φυστάμενοι φραγμοί δηλαδή τα προβλήματα που υπάρχουν με τα διάφορα πρότυπα προσβασιμότητας. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό σε εθνικό επίπεδο, καθώς τα κράτη θα καλούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις της συνθήκης, της σύμβασης. Συγγνώμη. Τώρα, πέραν αυτού, με αυτή την νομοθετική πράξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει την ευκαιρία να διευκρινίσει τι εστί προσβασιμότητα σε άλλα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος για τις δημόσιες προμήθειες ή σε πλαίσιο, παραδείγματος χάρη, όπως αυτό των υπηρεσιών από το ακουστικό τομέα. Έρχομαι στα ηθικά ζητήματα. Η έλλειψη παραδειγματο χαρη έχει ένα τίμημα. τομεα έχει κόστος η ελλειψη προσβασιμότητα εχει ενα μόνο, αλλά και η έλλειψη προσβασιμότητας. Το βλέπουμε αυτό και σε δύο υποθέσεις που συζητήθηκαν στην Αρμόδια Επιτροπή του Είχαμε την περίπτωση, την υπόθεση Νιουστή και Τάκασξ κατά Ουγγαρίας το 2013 και την υπόθεση Γιούγκελιν κατά Σουηδίας το 2014. Και έχουμε και άλλες δύο, επιθέσεις, δύο υποθέσεις αγγλικές. Δηλαδή χρειάζεται τα άτομα με αναπηρία να δίνουν τα στραπεζικά του στοιχεία, τον αριθμό πίν για τις ε, τραπεζικές του αλλαγές, Άρα να εμπιστεύονται. Και υπάρχει και το ενδεχόμενο της απάτη σε βάση αυτών των ατόμων. Δεν καλύπτονται και από τραπεζικά ασφαλιστικά ε, προγράμματα. Δηλαδή, αν έχουν δώσει το πιν τους αυτοί οι άνθρωποι σε κάποιον άλλο, οι τράπεζες τους ασφαλίζουν. Η περίπτωση, η δεύτερη της Σουηδίας, αφορά την απασχόληση και είναι κάτι πολύ σημαντικό ένα άτομο ε, με πρόβλημα όρασης δεν μπορούσε να προσληφθεί γιατί δεν είχε πρόσβαση στο σύστημα πληροφορικής μιας εταιρείας. Ενώ ήταν η καλύτερη για τη θέση, η συγκεκριμένη υποψήφια δεν μπόρεσε να πάρει τη θέση. Θεωρούμε λοιπόν ότι για αυτούς και για πάρα πολλούς άλλους λόγους θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει υπάρχει κοινωνικό, ε, συναισθηματικό ε, τίμημα, υπάρχει τίμημα σε ό,τι αφορά την υγεία και πλήττονται και τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι. Έχει την ε, ευκαιρία για αλλαγή ένωση με αυτή ακριβώς την νομοθετική πράξη για την προσβασιμότητα. Θα μπορούσε να ενισχυθεί ακόμη περισσότερη πρόταση, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε υπόψη ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο και θα πρέπει να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εμπειρογνώμονες για τις παρεμβάσεις τους. Εντάξει, ξεπεράστε τα πέντε λεπτά, να το πούμε και αυτό, αλλά δεν πειράζει. Τώρα, στο δεύτερο γύρο που θα ακολουθήσει τώρα θα μιλήσουν οι συγητές και οι συγητρίες. Ε, ο κύριος Άνταμ Κρόζα είναι ο συγητής για, για αυτό το θέμα. Άνταμ, σε παρακαλώ για δύο λεπτά ή Άνταμ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Θεωρώ ότι ο σκοπός της σημερινής ακρόασης είναι να ακούσουμε τις εμπειρογνώμονες, να ακούσουμε τις παρεμβάσεις τους και εμείς καθώς και οι σιώδεις εισηγητές ε, να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά που ακούσαμε στην έκθεσή μας. Θα ήθελα μόνο να βρίσκεται την προσοχή σας σε ένα σχόλιο, το οποίο μάλλον λείπει ένα σημείο, και δεν το εννοώ αρνητικά, όμως ε, υπάρχει μια μικρή παράληψη. Σε ό,τι ε, αφορά το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το με αναπηρία, ίσως να μην είναι εμπειρογνώμονες, έχουν όμως σημαντική εμπειρία. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να, να δώσουμε και το βήμα ε, και το λόγο σε αυτό το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για να μπορούν και εκείνοι να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώ περιμένουν από του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω να έχουμε εδώ ε, το χρόνο για αυτό ακριβώ το ζήτημα. Μετά προσβλέπω σε ε, συνεργασία με τους συναδέλφους, γιατί νομίζω ότι θα είναι μια πολύ χρήσιμη και ωφέλιμη εμπειρία. Όπως και να έχει, είναι μια μεγάλη πρόκληση όλο αυτό το εγχείρημα για μας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο. Ο κύριος Ρίτσαρτ Χάουιτ έχει το λόγο. Ο Ρίτσαρτ. Αλλά μάλλον ε, δεν ξέρω, δεν τον βλέπω. Δεν είναι στην αίθουσα. Helga Stevens, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εμείς βεβαίω ε, χαιρετίζουμε τη σημερινή ακρόαση. Είναι σημαντικό γιατί και τώρα έχουμε την, ευρύτερα την ευκαιρία ε, να συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό αυτόνομο σχέδιο ε, μαζί με τους εμπειρογνώμονες και Συμφωνώ με τον συνάδελφο Άνταμ ε, πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν και τα άτομα με αναπηρία και οι οργανώσεις τους, οι φορείς τους. Ε, θεωρώ ότι στις επόμενες συνεδριάσεις θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Γι' αυτό θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον χρόνο ομιλία μου και να τον ε, χαρίσω των εισαγωγικών στα άτομα ακριβώ από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Αν και εσείς συμφωνείτε. Ευχαριστώ. Äh. Πολύ ευγενικό αυτό εκ μέρου σα, Ingrid. Επόμενος, Μάριαν ε, Χάικιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις παρουσιάσεις. Λυπάμαι που δεν ήμουν εδώ εγκαίρως για να τις ακούσω όλες, όμως... Ε, έχω πολύ καλέ σημειώσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου όσοι έκαναν παρουσιάσει σήμερα. Είχαμε μια πολύ καλή εισαγωγή, Ελαφρώ διαφορετικέ οπτικέ γωνίες, το οποίο είναι θετικό γιατί πρέπει να δούμε το ζήτημα από όλε τι πλευρές. Εγώ, όπω και οι υπόλοιποι σκιώδεις ε, ανυπομονώ να συνεργαστώ με, με ε, στον τομέα. Σίγουρα δεν είμαι τόσο ειδήμων σε αυτά τα ζητήματα, έχω πολλά να μάθω. Όμω είμαι να ακούσω και ε, να αντιλήσω διδάγματα από την εμπειρία σε άλλες χώρες, γιατί έτσι μπορούμε, ελπίζω, να καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό κείμενο. Επομένω, συμφωνώ με τους υπόλοιπους ε, σκιώδεις εισηγητές. Θέλω λοιπόν και εγώ να συνεργαστώ με όλους αυτούς τους φορείς και να ε, καταλήξουμε σε ένα, μια πρόταση προσβασιμότητας που θα κάνει πραγματικά διαφορά στις ζωές αυτών των προσώπων. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να είναι στην αίθουσα η κυρία Κούνεβα. Η Τατιάνα έχει το λόγο. Η Τατιάνα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πάμε που μόλις ε, έφτασα ε, λόγω της αυξημένης κίνησης. Άκουσα ότι αναφέρθηκε η έλλειψη των εκπροσώπων ΜΚΟ για την ακρόαση και συμφωνώ απολύτως. Είναι σημαντικό να έχουμε εκπροσώπους ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων ατόμων με αναπηρία και εκπροσώπους άλλων φορέων σε αυτή την ακρόαση εφόσον η βασική αρχή σε αυτό το φάκελο ε, δεν είναι μόνο η τεχνική προσβασιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίε. αλλά και η κοινωνική διάσταση του ζητήματος. Και εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να κάνουμε ό,τι παίρνει από το χέρι μας ε, για να έχουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση και να σκεφτούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτά τα άτομα με αναπηρία για να αυξήσουμε την προσβασιμότητά τους ε, σε προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτά εν ολίγης από μένα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ούτε η Λάουρα Ατζέα είναι στην αίθουσα, ούτε και ο επόμενο ομιλητή. Ερωτώ λοιπόν. Ο Ντομινίκ Μαρτάν. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω ε, είναι πολύ σημαντική η σημερινή ακρόαση και χαιρετίζω όσου πήραν τον λόγο. Όμω, η πρόταση οδηγία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί ότι θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά και θα εξαλείψει τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία και θα διευκολύνει την συμπερίληψη και την ε, αυτονομία όλων ε, στην σημερινή κοινωνία. Όμως, με αυτή την ε, προσέγγιση και την προσέγγιση μάλλον ε, των προτύπων δεν κάνει ακριβώ αυτό. Δυσκολεύει τα πράγματα και για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί τίθεται και ζήτημα δημοσίων προμηθειών. Και έτσι φτάνω στο μεγάλο αλλά. Ενδεχομένω να φαίνεται ότι το θέμα αυτό της αναπηρίας κάπως το αξιοποιούμε για τους σκοπούς ε, της ε, ενιαίας αγοράς. Όμως, ε, για να αποδεχθούμε, θέλουμε εδώ να αποδεχθούμε την εναρμόνιση των αγορών και την ομογενοποίησή τους και έτσι πρέπει να κάνουμε την επιλογή μεταξύ της πρόσβασης σε, εμπόδι, συγγνώμη, σε εμπορεύματα και υπηρεσίες και αυτό οδηγεί σε σύγχυση η επικύρωση τη ε, Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτα απ' όλα, θα μπορούσε να αποτελέσει δούριο ύπο για να επιβάλλουμε ε, την ενιαία αγορά και μια φεντεραλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. So, Πολύ ωραία. Έχω λοιπόν την ε, εξή πρόταση. Έχω στον κατάλογο μου άλλα δύο μέλη και μετά θέλω να ρωτήσω. Ε, συμφωνείτε με αυτά που πρότειναν οι Σνάλφοι Κόζαν Στίβεν Νόρτον, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ ε, Αναπηρίας, ε, να μιλήσει δηλαδή αυτή η κυρία για δύο λεπτά. Και αφού μιλήσει εκείνη, μετά θα μιλήσει ο συγητής και κλείνει κατά τα άλλα ο κατάλογος. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Εγώ είμαι από το φόρουμ, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας. Το φόρουμ μας ε, εκπροσωπεί μέλη με αναπηρία και για πάρα πολλά χρόνια ήμασταν οι πιο διαπρίσιοι υποστηρικτές ε, της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο και ευχαριστώ και τα άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, σκέπτονται κυρίως τις υποχρώσεις που έχουν ε, με βάση τις συμβάσεις υποχρώσεις να δραστηριοποιηθούν για άτομα με αναπηρία. Η νομοθεσία περί αναπηρίας είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την καθημερινή ζωή πάρα πολλών ανθρώπων με αναπηρία όπως επίσης και τη ζωή 190 εκατομμυρίων ηλικιωμένων ατόμων στην Ευρώπη. Εάν λοιπόν εγκριθεί και εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία αυτή θα μπορούν τα άτομα με αναπηρία να αγοράζουν ε, ηλεκτρονικά και να κάνουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όμως ε, για να είναι αποτελεσματική νομοθεσία ε, πρέπει να διευρυνθεί το πλαίσιο εφαρμογή της και αυτό σημαίνει ότι θα χαρούμε πάρα πολύ να συνεργαστούμε με τα μέλη της Επιτροπής. Οι περισσότεροι θα συμφωνούν ότι τα ATM ε, πρέπει να είναι προσβάσιμα και σε άτομα με αναπηρία ε, Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ ευτυχείς ε, που ακούσαμε και τις ε, παρεμβάσεις των εμπειρογνωμών που ζήτησαν να διευρυνθεί ε, η εμβέλεια αυτή τη νομοθεσία βεβαίω και πρέπει να υπάρχει ένα μηχανισμό εφαρμογή και ακούσαμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα ουσιαστικό τέτοιο ε, μηχανισμό. Κατά τα άλλα, πάρα πολλέ εξαιρεσει ε, μπορούν να αποδυναμώσουν το κείμενο, γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύ προσεκτικά. Ελπίζουμε η Επιτροπή επασχόληση να τα έχει όλα αυτά κατά νου και τελικά θα έχουμε ε, μια νομοθεσία αντάξια στην, στο όνομά της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ε, τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Κοιτάξτε, όταν ε, δίνω το λόγο στην εισηγήτρια και δεν είναι παρούσα, να μας λένε αμέσω οι πολιτικές ομάδες ε, ποιο την αντικαθιστά. Γι' αυτό το λόγο έχει τώρα η κυρία Γιούτα Στάνρουκ εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Μάλλον δεν με είδατε προηγουμένως που ζήτησα το λόγο. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπήρων και Αναπηρίας ε, είχε τη δυνατότητα να λάβει το λόγο. Ο εισηγητής ε, δεν το είχε προτείνει αυτό στον κατάλογο των ομιλητών. Εμείς το είχαμε συζητήσει στις συνεδρίες των συντονιστών. Είχαν διαφωνήσει περισσότεροι, αλλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είχατε τη δυνατότητα να λάβετε το λόγο, γιατί πιστεύω δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για άνθρωπα, αλλά και με τους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ακρόαση λοιπόν κατέδειξε ότι έχουμε ακόμα να κάνουμε πάρα πολλά, γιατί το θέμα δεν είναι να καταπολεμάμε και αντιμετωπίζουμε αντικά την κοινή αγορά, γιατί ξέρετε τα άτομα με αναπηρία εξαρτώνται από το να παίρνουν τα κατάλληλα προϊόντα, απαραίτητα από την πατρίδα τους, αλλά κυρίως ευρύτερα από την κοινή αγορά. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη είναι ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μπλοκάρει την οριζόντια οδηγία ε, που αφορά στην κατάργηση των διακρίσεων. Αν δεν ίσχυε αυτό θα προχωράγαμε πολύ γρηγορότερα. Ε, στο Κοινοβούλιο νομίζω έχουμε ήδη προχωρήσει. Τα βασικά προβλήματα είναι η πρόσβαση σε κατάλληλη στέγαση, σε ε, σε πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τα άτομα με αναπηρία. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που γίνεται και θεωρώ ότι αν έχετε και κάποια άλλα πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα όπου να μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Επιτροπής, αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό. Το παράδειγμα που είπατε με τα ETM, αυτό το αναφέρατε συχνά και αυτό είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα για να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε βελτιώσεις. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Αν μπορείτε και τα παραδείγματα μάλιστα να μας τα δώσετε και σε γραπτή μορφή, αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο για την περαιτέρω διαδικασία. Άννα ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους όσοι συμμετέχουν στη συζήτηση. Σήμερα συζητάμε για την πρόταση της Επιτροπής ε, ε, προσαρμογής ε, των διοικητικών ε, προδιαγραφών για προϊόντα και υπηρεσίες. Είμαι λοιπόν ε, αισιόδοξο ότι θα κατορθώσουμε υπό την καθοδήγηση του κ. Κόζα να βρούμε σημαντικές και ουσιαστικές λύσεις. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάποιες λεπτομέρειες. Το ζητήσατε και θεωρώ ότι υπάρξουν αρκετές προσθήκες, γιατί δύο πράγματα είναι σημαντικά για μένα τουλάχιστον. Πρώτον, να γίνει, να υπάρξει αναγνώριση σε όλη την Ευρώπη των σκυλιών για τυφλούς και κοφούς. Ε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται συχνά λόγος για ανθρώπους που εξαρτώνται πλήρως από τα σκυλιά συνοδούς. Όμως τα σκυλιά αυτά ε, τα βρίζουν και τα πετάνε και έξω μάλιστα από εστιατόρια και από άλλους δημόσιους χώρους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για αυτά τα σκυλιά σύνοδους και θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα παντού. Είναι ευπρόσδεκτα τα σκυλιά σύνοδοι. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι σημαντικό για μένα είναι το εξής. Ίσως βέβαια αυτό λιγάκι δημιουργήσει κάποια σύγχυση, όμως να υπάρχει παντού στην Ευρώπη το δικαίωμα θυλασμού. Γιατί βλέπουμε ε, σε πολλές περιπτώσεις γυναίκες οι οποίες πάνε στα καφενεία, πάνε στα πάρκα, πάνε στα μαγαζιά, στα τρένα, ε, θέλουν να θυλάσουν και τις πετάνε έξω. Τις πετάνε γιατί θυλάζουν τα μωρά τους. Μα αυτό είναι διακριτική μεταχείριση. Ο αποκλεισμό ε, λοιπόν παροχής υπηρεσιών στην κοινή αγορά, αυτό είναι κάτι που θίγει πάρα πολλές μητέρες οι οποίες θα ήταν ε, όλες πολύ ευχαριστημένες αν μπορούσαμε να τους ε, εγγυηθούμε σε ολόκληρη την Ευρώπη το δικαίωμα θυλασμού και σε δημόσιους χώρους. Ε, μην ξεχνάμε ότι ε, στη Βρετανία υπάρχει τέτοια νομοθεσία που απαγορεύει διακριτική μεταχείριση εις βάρος των θύλαζουσών γυναικών. Και νομίζω ότι έχουμε τις αρμοδιότητες για να τα πετύχουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά πρέπει να μου το εξηγήσετε λιγάκι. Εγώ δεν ήξερα ότι ο θυλασμός έχει σχέση με την αναπηρία, ότι η αναπηρία τέλο πάντων. αν θα τα πούμε αυτά μετά. Τώρα ο εισηγητή έχει το λόγο. Παρακαλώ. Kedves kollégák, köszönöm a hozzászólásokat is. Nem tudom, hogy az én... Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχω τα εξή ε, σχόλια, καθώς θα κλείσουμε αυτό το σημείο της μέσα διάταξης. Ήθελα μόνο να πω ότι ε, στην αρχή είχα πει ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο και στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Πολλές φορές όμως ε, ακούσαμε ότι το πεδίο εφαρμογή είναι εξαιρετικά στενό Κατά τη γνώμη μου, το ρέτο που είναι το εξή. Εάν η νομοθετική πρόταση αυτή τη στιγμή ε, δεν θεσπίσει ορισμένες αρχές, τότε πώς θα καταφέρουμε τα άτομα με αναπηρία να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες. Άκουσα τους συναδέλφους και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που εφήγει περισσότερο. Αυτό θα είναι το μεγάλο μας καθήκον να φροντίσουμε, να μην περιορίζονται οι ε, απαιτήσει αυτές, τα προϊόντα και υπηρεσίες να είναι προσβάσιμα σε όλους και παντού. Σε σχέση τώρα με τα σχόλια του Γάλλου συναδέλφου, θα ήθελα να πω το εξής. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να συγχέουμε και να μπερδεύουμε τα ε, δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία με εθνικά εγχώρια ζητήματα. Και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, ε, για σήμερα τουλάχιστον τελειώσαμε αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να παρακαλέσω τους ε, εμπειρογνώμονες ε, να μας καταθέσουν προτάσεις συμπληρωματικές έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας και θα ήθελα να επισημάνω ότι με τη βοήθεια των διερμηνέων της ε, νοηματικής ε, και των ε, διαφανειών αυτών που είναι κάποιος από το Αμβούργο που δεν τουρίζουμε καν. Κατορθώσαμε να έχουμε μια πολύ καλή συζήτηση. Στις 20 Οκτωβρίου θα υπάρχει ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες. Στις 29 ψηφοφορία και 25-26 Ιανουαρίου θα συζητήσουμε στην Ολομέλη του 17 προφανώς. Πολύ ωραία. Πάει αυτό το θέμα. Πάμε στο επόμενο. Επόμενο θέμα είναι ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η Συγεία η Μαρία Ζωάου Ροντρίγκες που σήμερα δεν θα την ξεχάσω όπως την ξέχασα την προηγούμενη φορά θα είμαι προσεκτικός. Καλωσορίζω τον Άλαν Λάρσεν, τον ειδικό εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον κύριο Γιούγκα, ο οποίος έχει έρθει σήμερα κοντά μας. Ε, σας είπα ε, να το ξαναπώ μάλλον, επειδή υπήρξαν κάποιοι που καθυστέρησαν να έρθουν, ε, έχουμε χρόνο αγόρευση σε δύο λεπτά και για την Μαρία και για τον Τσάο και μετά ο κύριος Λάρσον. Ε, θα μπορεί όμως εκείνος να μιλήσει για δέκα λεπτά, γιατί εκείνος είναι εξωτερικός εμπειρογνώμονας και γι' αυτόν δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Η Μαρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που ξεκινώ με την παρουσία αυτών των συναδέλφων το έργο πάνω σε αυτή την έκθεση. Θέλω με τη βοήθεια όλων να έχουμε μία έκθεση σημαντική με νόημα γιατί νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός πυλώνας ε, κοινωνικών δικαιωμάτων που θα ανταποκρίνεται στι ανησυχίες των πολιτών ε, για να μπορέσουν να κτίσουν έλεγχο τη κατάστασης και για να Υπάρχει μια επανεξισορρόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Ευρωζώνης. Θέλω να καλωσορίσω τις προτάσεις της Κομισιόν. Βλέπω βέβαια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω σε αυτές τις προτάσεις πρέπει να οικοδομήσει και να πάει πιο μακριά ακόμα με στόχο μια δεσμευτική συμφωνία ή δυνατόν μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων όμω. Η δεσμευτική συμφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται και από έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή, την υλοποίηση του πυλών αυτού. Ζητούμε, όσο αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα, γενναίες ιδέες, τολμηρές ιδέες, ιδίως ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. αυτή η εγγύηση για την ολιά. Πρέπει να γίνει ένα νέο δικαίωμα, για παράδειγμα, ιδίω ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Οι γυναίκες επίσης θα πρέπει να ενισχυθούν. Θα πρέπει να δούμε τι άδειε ε, δίνονται και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα διάφορα προγράμματα και ακόμη οι συνθήκε εργασία θα πρέπει να είναι εξωπρεπεί και δίκε. και αυτό να είναι εγγυημένο για όλου του εργαζομένου ανεξαρτήτω μορφή απασχόληση. Θα πρέπει επίση θα πρέπει να έχουμε υπόψη και την ψηφιακή επανάσταση που συντελείται αυτή την εποχή και τι επιπτώσει έχει. Γι' αυτό και προτείνουμε να υπάρχει οδηγία η οποία θα καθορίζει δίκαιους όρου για όλε τις μορφές απασχόλησης. Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους κοινωνικούς κινδύνους. Θέλουμε μια εγγύηση για τα παιδιά. Έχουμε την εγγύηση για την νεολαία. Όμως πρέπει να δούμε και τα προβλήματα των εργαζόμενων φτωχών. Και θέλουμε και ένα πλαίσιο για την καθιέρωση ελάχιστου εισοδήματος, κατώτατου εισοδήματος. Και τα, το συνταξιοδοτικό είναι ένα ζήτημα. Η βιωσιμότητα σίγουρα εξαρτάται από την ενεργογύρανση, το ξέρουμε αυτό. Όμως δεν υπάρχει καλύτερος α, τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα από την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης παντού. Επίσης θα πρέπει να έχουμε αξιόπιστα μέσα. Και αυτό σημαίνει νομοθεσία αλλά και επανεξισορρόπηση της οικονομικής διακυβέρνησης. Δηλαδή, πολύ περισσότερη προσοχή πρέπει να δώσουμε σε κοινωνικούς δείκτες. Προτείνω να έχουμε έναν ε, κώδικα σύγκλησης, αν θέλετε, ώστε να υπάρχει μακροοικονομική εποπτεία. Και όταν ανακύπτουν μεγάλες ανισορροπίες κοινωνικά προβλήματα, να μπορεί να ενεργοποιείται η δράση και να ε, δίνονται περισσότερα μέσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και όταν μιλώ για περισσότερα μέσα, εννοώ και οικονομικά. Για τη στήριξη των κοινωνικών επενδύσεων πρώτα απ' όλα. Να υπάρχει σχετικό κανόνα ε, στην ε, διαδικασία δημοσιονομική προσαρμογή. Βέβαια, πολλά εξαρτώνται και από τη δυνατότητά μα να αντιμετωπίσουμε την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Διότι εκεί εντοπίζουμε σημαντικές πηγές εσόδων Και βέβαια θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα. Έχουμε το Ευρωπαϊκό, Στρατη... το Ευρωπαϊκό Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα πρέπει να εστιάζει πολύ περισσότερο στην δημιουργία καλών θέσεων εργασία και κοινωνικών επενδύσεων. Έχουμε όμως και τα διορθωτικά ταμεία, που είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την κοινωνική συνοχή τέλος. Υπάρχουν και ειδικέ ανάγκες της Ευρωζώνης. Εδώ προτείνω ένα μέσο σύγκλησης και την αντιμετώπιση των ασυμμετρικών κραδασμών. Εμείς εκπροσωπούμε του πολίτες και πρέπει να είμαστε τολμηροί για να μην είμαστε κάτω από τις προσδοκίες που έχουν ε, να αποθέσει και ελπίδες που έχουν να αποθέσει οι πολίτες σε εμάς. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Λάρσον λοιπόν, ο οποίος είναι ειδικό εμπειρογνώμονας ε, απεσταλμένος του κύριου Γιούγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλό απόγευμα. Είναι μεγάλη μου χαρά ε, να παρουσιάζω εδώ τις συνεχιζόμενες ε, διαβουλεύσεις κατόπιν ε, πρωτοβουλίας του κυρίου Γιούγκερ για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Μιλούμε εδώ για την απασχόληση, τα κοινωνικά δικαιώματα στην εργασία και κοινωνική δικαιοσύνη και ασφάλεια. πρέπει εγώ να λειτουργήσω ως ε, σύμβουλος και όχι ως εκπρόσωπος τύπου. Γι' αυτό και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ να ακούσω και τις δικές σας ε, συμβουλές και να συμμετάσχω στις ε, εργασίες για την έκθεση αυτή το θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Πυλώνα είναι προτεραιότητα της Επιτροπής Juncker, όπως είχε τεθεί το 2014 και, και μάλλον εστιαζόμαστε στην απασχόληση και την κοινωνική συμπερίληψη. Το 2016 ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και ο πρόεδρος Γιούνκερ επιβεβαίωσε αυτό το μήνυμα και στην ε, ομιλία του ε, πριν από δύο εβδομάδες, ε, όπου έλεγε τα τελευταία τρία χρόνια 8 εκατομμύρια ακόμη άνθρωποι έχουν βρει μια θέση απασχόληση, όμω η ενεργεία παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, καθώ και κοινωνική αδικία και ανισότητα. Γι' αυτό και θα πρέπει τάχιστα να εργαστούμε πάνω στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, γιατί η Ευρώπη δεν είναι αρκετά κοινωνική. Αυτό ήταν το μήνυμά του. Αυτό, εν συντομία, είναι το πολιτικό υπόβαθρο πίσω από την πρωτοβουλία Juncker. Τώρα θα ήθελα να στραφώ στο οικονομικό κοινωνικό και δημογραφικό πλαίσιο και προκλήσεις που ε, στοχεύει να αντιμετωπίσει αυτή η πρωτοβουλία. Στο έγγραφο διαβούλευση έχουμε τέσσερι πολύ καλού λόγου για μια νέα αρχή για την κοινωνική Ευρώπη. Πρώτον, έχουμε μακρόπνοε επιπτώσει τη οικονομική κρίση που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια σε ό,τι αφορά την χαμηλή ανάπτυξη, την ε, ανεργία, την ένδυα, του κοινωνικού αποκλεισμού. με τις ε, αλλαγές στη νέα ψηφιακή οικονομία, όλα αυτά αλλάζουν και τον, ε, ε, την οικονομία μας, την αγορά μας. Μπαίνει στο πλαίσιο και η ψηφιακή οικονομία, η ψηφιακή αγορά. Πρέπει έτσι να έχουμε και εμείς επίγνωση των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν. Τρίτον, δημογραφικές και κοινωνιακές τάσεις, κυρίως ό,τι αφορά την γυράσκουσα Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις εργαζόμενους για κάθε ηλικιωμένο. Στην επόμενη γενιά θα έχουμε μόλις δύο ε, εργαζόμενους για κάθε συνταξιούχο. Έτσι, το κοινωνικό μα συμβόλαιο τίθεται υπό σημαντική πίεση. Και τέταρτον, η σημασία των αποκλήσεων αντί τη σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών, ε, ιδίω ό,τι αφορά την Ευρωζώνη. Οι κακές επιδόσεις μετά την κρίση και οι τεράστιες προκλήσεις ενώπιών μας μας οδηγεί στο ερώτημα να εξετάσουμε τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί στην κοινωνική Ευρώπη. Που είναι η άβολη ερώτηση, όπως την αποκαλώ εγώ, και είναι η εξή. Πώς γίνεται η ανέχεια και οι ανισότητες να είναι τόσο ευρέως στην Ευρώπη, παρότι έχουμε τα καλύτερα κοινωνικά συστήματα στον κόσμο και παρότι έχουμε την πλέον εύρωστη αγορά στον κόσμο με 500 εκατομμύρια ε, πολίτες και τόσες επιχειρήσεις. Είναι το πρόβλημα για δυναμία στην εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων, μεγάλα ε, κενά στο δίκτυο ασφαλείας ή άλλοι λόγοι. Στην διαδικασία διαβούλευση θα πρέπει να θίξουμε αυτά τα ερωτήματα και να βρούμε και απαντήσει. Ιδάλω δεν θα είμαστε σε θέση να ε, προσδιορίσουμε το απαραίτητο πακέτο μεταρρύθμιση. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται συχνά στη διαβούλευση αυτή είναι ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ε, σημερινού ε, κοινωνικού εκτιμένου και του νέου πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα. Η απάντηση που δίνω είναι ότι το υφιστάμενο κοινωνικό ε, και εκτιμένο ε, αφορά συγκεκριμένα βήματα που έχουμε κάνει, σιγά σιγά τα έχουμε συζητήσει και με μια πολιτική διαδικασία καταλήγουμε σε λύσεις. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων διαφέρει. Χρειαζόμαστε μια πιο ληστική προσέγγιση που θα συμπεριλαμβάνει και καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών και κοινωνικών εξελίξεων την τελευταία δεκαετία, αλλά και των προκλήσεων που έχουμε ενώπιόν μας. Ε, την γυράσκουσα Ευρώπη και τις αποκλήσεις. Είναι πολύ πιο ε, σημαντικό το εγχείρημα και δύσκολο να επιτευχθεί, όμως κάποιος θα πρέπει να το κάνει. Μπορούμε να βασιστούμε σε μία αναδυόμενη παγκόσμια συνένεση ε, και κοινή κατανόηση για τον ρόλο της κοινωνικής πολιτικής. Ένα από ένα στοιχείο είναι τα συμπεράσματα του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του ΟΣΑ ε, και του Διεθνού Γραφείου Εργασία, για τι αυξανόμενε ανισότητε, που δεν είναι μόνο κοινωνικό πρόβλημα, αλλά και οικονομικό μάλλον πρόβλημα. Οι αυξανόμενες ανισότητες αποτελούν εμπόδιο ε, στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτό ήταν το μήνυμα αυτών των διεθνών ε, οργανισμών ε, για την συνάντηση πέρσι του G7. Είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει επαναληφθεί πολλές φορές, κυρίως από την κυρία την επικεφαλής του Διεθνούς ομοσπονδικού Ταμείου, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον κύριο Ντράκη. Πρέπει εδώ στο έγγραφο διαβούλευσης να συμπεριλάβουμε και ένα μήνυμα για την κοινωνική πολιτική ως παραγωγικό παράγοντα βάσει της παρατήρησης ότι τα κράτη-μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις είναι και τα κράτη-μέλη με το πλέον προηγμένο και καλά σχεδιασμένο κοινωνικό σύστημα. Το τρίτο αφορά την ευελιξία και ασφάλεια. Είναι στοιχεία που αλληλοσυμπληρώνονται, δεν αλληλοποκλείονται αυτά τα δύο. Όμως ε, θα πρέπει να ανασχεδιάσουμε την κοινωνική ε, προστασία σε μια ευέλικτη οικονομία πλέον. Και έχουμε βεβαίως και τις ανισότητες ε, της έμφυλες. Πρέπει να διασφαλίσουμε τις ίσες ευκαιρίες ε, για όλους, κάτι το οποίο αποτελεί μεγάλη πρόκληση για μας. Τώρα, πώς ε, διαρθρώνεται αυτή η διαδικασία διαβούλευσης. Αρχικά έχουμε το υφιστάμενο και εκτιμένο, τι πάει καλά και τι όχι. Μετά για το μέλλον εξετάζουμε το μέλλον λοιπόν της απασχόλησης και των ε, συστημάτων πρόνοιας. Και μετά έχουμε και τον κοινωνικό πυλώνα ε, στο πλαίσιο της ΟΝΕ. Θέλουμε λοιπόν να θέσουμε θεματολόγιο, να αυξήσουμε τις γνώσεις μας και να θεσπίσουμε πολιτική και προσθέτω εδώ ορισμένες ε, σκέψεις ε, για τις μελλοντικέ μας ε, συνεδριάσεις. Έχω συμμετάσχει σε πολλές τέτοιες συναντήσεις εδώ στις Βρυξέλλες, επιμέρους επιτροπές, συναντήσεις με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά και στα κρατημέλη, Βερολίνο, Βιέννη, Ρώμη, Χάγη, Κοπενχάγη και Ναμύρ το Φθινόπορο. Από αυτές τις συζητήσεις θα ήθελα να αναφέρω μόνο μερικά στοιχεία. Πρώτον, αυτό που αποκαλώ μαύρη τρύπα των ευρωπαϊκών κοινωνικών συστημάτων. Είναι μία έλλειψη γεφυρών ε, που οδηγούν κάποιον πάλι πίσω στην αγορά εργασία. Οι πολιτικές κρατών μελών δεν είναι καλά σχεδιασμένες για την δυναμική μετάβαση που ε, παρατηρείται στις ε, ευρωπαϊκές αγορές. Είναι θέμα σχεδιασμού και καλύτερη αξιοποίηση πόρων. Τα δικά μας συστήματα ε, είναι προσαρμοσμένα στις αγορές εργασίας ε, του παρελθόντος με επιδόματα ανεργίας αλλά πολύ λίγες ε, διεξόδους και γέφυρες για να επανέλθει κάποιος στην αγορά εργασίας. Τα στατιστικά δείχνουν ότι κατά πέντε όρο 10% των ανέργων έχουν προσφορές για μια νέα κατάρτιση ή κάτι άλλο. Το 90% όμως βλέπουμε ότι καλούνται να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας χωρί καθόλου δεξιότητε ή με τι παλιέ του δεξιότητε. Και αυτό αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη νέα οικονομία. Αυτό αποκαλώ εγώ μαύρη τρύπα ε, των ευρωπαϊκών κοινωνικών μα συστημάτων. Και αυτό είναι το πλέον πιαστικό ζήτημα στην ε, προετοιμασία ενό ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Δεύτερο στοιχείο, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις μαύρες τρύπες, είναι η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Εδώ αυτό συνδέεται και ε, τις παραδοσιακές μορφές ε, συμβάσεων απασχόλησης που πλέον υπονομεύονται και αντικαθίστανται από νέες ε, μορφές. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να σταματήσουμε βεβαίω τις τεχνολογικές εξελίξεις. Πάντα τεχνολογία θα υπερνικά ε, τη, τη δημόσια πολιτική. Χρειάζεται λοιπόν καινοτομία και από την άλλη πλευρά του νομικού πλαισίου για να παρέχεται ασφάλεια στους εργαζομένους ενώ θα επιτρέπουμε και νέες ευέλικτε μορφές οργάνωσης της απασχόληση. Τρίτο ερώτημα, το οποίο τίθεται συχνά στη δικαστική διαβούλευση, είναι πώ ο Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα ενταχθεί στι μακροοικονομικέ πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών μελών. Επισήμω, μπορώ να σα πω ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο διαβούλευση, όμω εντάσσεται στο τρίτο πεδίο, τρίτη φάση ε, των ε, διαδικασιών και το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πιστική ε, μακρο, μακροοικονομική πολιτική στρατηγική γιατί αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Τέλος, τι θα κάνει ο καθένας, περισσότερη Ευρώπη ή περισσότερες ευθύνες για τα κρατη Γεγονό είναι ότι τα κράτη-μέλη έχουν την αρμοδιότητα για την αγορά εργασία και την κοινωνική πολιτική και θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με του κοινωνικού εταίρου. Ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να θέσει το ζήτημα επιτάπητο, να θέσει τα πρότυπα ε, και να τεθεί επικεφαλή για να εξευρεθεί μια νέα ισορροπία μεταξύ τη οικονομική και τη κοινωνική Ευρώπη, όπω έχουν ζητήσει πολλοί. Πιο πρόσφατα από τους ε, αρχηγούς των κυβερνήσεων, αλλά και από τους επικεφαλείς ε, Δουνουτού και ΕΚΤ. Σε μερικού μήνε, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει τη νέα τη πρόταση για το νέο κοινωνικό σύστημα τη Ευρώπη και θα παρουσιάσει ένα νέο ληστικό όραμα για το μελλοντικό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Να υπογραμμίσω ακόμα ένα στοιχείο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην πεπατημένη. Τα παλαιά μοντέλα πλέον δεν μας κάνουν. Η οικονομική ανάκαμψη είναι ανεμική και έτσι δεν επαρκεί αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται να λειτουργήσουμε μόνο με μικρές αλλαγές δεξιά και αριστερά. Πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη και την απασχόληση και φιλική προς, το, προς τους επιχειρήσεις, αλλά και πιο κοινωνική. Τα τελευταία δέκα χρόνια ούτε φιλική προς τις επιχειρήσεις ήμασταν, ούτε κοινωνική. Πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε και τα δύο. Με αυτά θα κλείσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, με ενδιαφέρον θα παρακολουθώ τις εργασίες σας και θα διαβάσω την έκθεση όταν ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λάρσεν. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε τώρα με τους σκιώδης ηγητές. Δύο λεπτά έκαστος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ροντρίγκη, την εισηγήτρια, για το κείμενό τη. Ο Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων δεν πρέπει να μείνει μόνο σε μια δήλωση καλών προθέσεων και συμφωνώ πλήρω με αυτό. Μπορούμε να μιλήσουμε ε, για μέρε για ε, αυτό το ζήτημα, όμω έχει έρθει η ώρα να περάσουμε στην πράξη, σε μία ακρόαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά και σήμερα η συγγήτρια αναφέρει ότι μπορεί να υπάρξει αυτό ο πυλώνας από νέα ή αναθεωρημένη νομοθεσία, από μηχανισμού ε, διαμόρφωσης πολιτικής, αλλά και από οικονομικού μηχανισμού. Θεωρεί ότι με αυτά ακριβώ τα στοιχεία μπορούμε να προχωρήσουμε και να μεριμνήσουμε, ούτω ώστε να είμαστε έτοιμοι και για το μέλλον, σε έναν κόσμο που αυξάνονται οι αλλά και που ε, αλλάζει συνεχώς ο ορισμός της απασχόλησης, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος προηγουμένως. Θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε, αλλά και τι μπορούμε να πετύχουμε. Σε μια εποχή όπου τα αρνητικά ε, συναισθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάρει το πάνω χέρι πλέον σε ορισμένε χώρες, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, τι ακριβώς θα κάνουμε. Αν θα διαμορφώσουμε νέες δομές, εγώ θα έλεγα όχι, να ενισχύσουμε τις εφιστάμενες δομές. Πρέπει όμω να δούμε και τι θα καταργήσουμε προκειμένου να αυξήσουμε και πάλι την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτέ τι τρει κατηγορίε που αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, ίσε ευκαιρίε στην πρόσβαση στην αγορά εργασία, ε, δίκαιοι όροι απασχόληση και ε, επαρκές ε, πλαίσιο κοινωνικής προστασίας. Και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να έχουμε μια φιλόδοξη έκθεση σε αυτό το πεδίο. Η συγγήτρια έχει ζητήσει να είμαστε τολμηροί και συμφωνώ απολύτως. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και πραγματικά προσβλέπω στη συνεργασία με την κυρία Ροντρίγκες. Πολύ ωραία. Εκ μέρους ε, του ECR παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. και ε, σκιώδης ηγητές ε, της ε, ομάδας μου χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να συμμετέχω και εγώ στη σημερινή συζήτηση για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα και ευχαριστώ τον Τιον Λάρσεν. Γνωρίζετε το όραμα που εξέφρασε κάποιος το 2004. Γνωρίζω ότι αυτό το όραμα πια δεν ισχύει, αλλά εμένα μου αρέσει. Αναφέρει λοιπόν ο συγγραφέας ότι ονειρεύεται μια Ευρώπη όπου εκτός από το άτομο θα υπάρχει και η κοινωνία και θα υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και όχι ανταγωνισμός. Ε, θα προηγείται η ποιότητα του κέρδους ε, στην κοινωνία, θα υπάρχουν οικογενειακές σχέσεις. Δηλαδή το ε, παλιό αμερικανικό όραμα του self-made αυτό έχει μετατραπεί σε όραμα του Τραμπ. Σήμερα εγώ θεωρώ ότι η Ευρώπη τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά με τις ε, κοινωνικές της ιδέες. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε. Ε, θα τις ε, υλοποιήσουμε αυτές τις ιδέες στο μέλλον. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε στο πλαίσιο του κοινωνικού πυλώνα. Και η Κομισιόν, όπως ξέρουμε, μέχρι το Δεκέμβρη καλεί όλους τους πολίτες και όλους άμεσα ενδιαφερόμενες για ε, διαπραγματεύσεις. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ένα τμήμα μιας πραγματικής bitter regulation και εμείς, αν ε, στο Κοινοβούλιο δεσμευτούμε πολύ νωρίς, νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Ε, συζητάμε για το ε, πώς θα πρέπει να είναι τελικά αυτός ο πυλώνας, αλλά ας προσπαθήσουμε να εγγυηθούμε υπεραξία. Εγώ αυτό ακριβώς εύχομαι να προκύψει από τις συζητήσεις για τον κοινωνικό πυλώνα και εμείς αυτά θα πράξουμε ως ECR. Εκ μέρους των ε, φιλελευθέρων, παρακαλώ για δύο λεπτά. Ενρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πολύ πλοκό το θέμα. Τι να πω μέσα σε δύο λεπτά, μόνο τα πιο σημαντικά, δηλαδή να ευχαριστήσω την εισηγητρία για τη δουλειά που έχει ήδη κάνει και να πω ότι η ομάδα Άλντε φυσικά και θεωρούμε ότι θα πρέπει να πέφτει το άρθρο αλλά σημαντικό επίσης θεωρούμε αυτή τη στιγμή όπως είναι τα πράγματα και είπε και από το ΕΛΚ, να δώσουμε κοινωνική διάσταση στην Ένωση. Η Ευρώπη δηλαδή δεν είναι απλά ένα σύστημα δημιουργίας ενίων νομισμάτων και οικονομίας, αλλά είναι και ένα σύστημα που ανησυχεί και ασχολείται και με την ευημερία των ανθρώπων και με τα ανθρώπινα και κοινωνικά τους δικαιώματα. Γι' αυτό θέλουμε να το στηρίξουμε, το εγχείρημα αυτό. Και υπάρχουν πολλά σημεία της έκθεσης με τα οποία συμφωνούμε. Μου, λείπει ένα, μου μένει ένα λεπτό και δεν θα το δαπανίσω για να μιλάω για τα ρόδινα της κατάστασης, αλλά για τις άλλες πτυχές. Ε, παίρνουμε μεγάλη απόσταση από όλα αυτά τα ποσοτικά. 30%, 70%. Θέλω να αποφεύγουμε τα ποσοστά, γιατί πολλές φορές ε, χρησιμοποιούμε παράλογα μαθηματικά, ε, μιλάμε για κάποιους μέσους όρους, φτάνουμε εκεί και μετά αυτό δημιουργείται ένας άλλος μέσος όρος και ούτω καθεξής. Θέλουμε ε, να μην επιβάλλουμε ένα κοινωνικό μοντέλο ενιαίο, αλλά να μιλάμε για αυτή την κοινωνική οικονομία της αγοράς, που την αναφέρουν και συνθήκε. συνθήκες. Αλλά ενιαίο μοντέλο είναι δύσκολο όταν έχουμε 28 διαφορετικά. 27, συγγνώμη τώρα, 27 μείναμε. Και θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με τις διάφορες μορφές σύμβασης και τι μεταχείριση θα έχουν. Όταν μπούμε στα συγκεκριμένα λοιπόν και ιδίως στα βραχυπρόθεσμα μέτρα, εκεί θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή πλατφόρμα συζήτηση. Δυσκολίες θα υπάρχουν πάντω, θέλω να το πω. Επίσης, υπάρχουν κάποιες προτάσεις που δεν περιλαμβάνονται, που θα θέλαμε να μπουν. Ε, για, θα μπορέσουμε να σας τα γράψουμε στη συνέχεια ε, σε τροπολογίες και έτσι θα βοηθήσουμε, πιστεύω, την εξαιρετική μας συζήτηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκάμπιτσιμα εκ μέρου τη ΓΚΟΕ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάρσον και τον συνάδελφο Ροντρίγκε για τι ε, παρεμβάσεις του και την κυρία Ροντρίγκε, με την οποία συμφωνώ απόλυτα γιατί είπε εκείνη ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένες προτάσεις, εργαλεία, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες δυνατότητες χρηματοδότησης έτσι ώστε πραγματικά να οικοδομήσουμε μια κοινωνική Ευρώπη. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάπως τα πρότυπα γιατί μιλάμε συνέχεια για τέσσερις βασικές πολιτικές ελευθερίες, αλλά αυτές οι ελευθερίες ε, υποτάσσονται στην προστασία, στην πραγματική προστασία της εργασίας και έτσι δεν μπορεί να ανανεωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ενταρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρότι εσείς κύριε Λάρσον λέτε ότι ε, δεν ανήκετε στην Κομισιόν αλλά είστε σύμβουλος, σας παρακαλώ να έχετε κατά νου ότι η Κομισιόν οφείλει να καταθέσει μια πρόταση που να είναι πιο συγκεκριμένη από αυτά που έχουμε διαβάσει. Πάρα πολύ γενικά αυτά, δηλώσεις προθέσεων. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι όταν μιλάμε για συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την ε, Κομισιόν πρέπει να υποβάλουμε κάτι το οποίο να είναι συγκεκριμένο, όχι να υπόσχεται χωριά του Ποτέμκιν, αλλά να ε, πείθει τους ανθρώπους ότι μπορούν να εργαστούν πραγματικά από την εργασία τους και όλοι οι άλλοι ότι θα μπορούν να ζουν, να ζουν αξιοπρεπώς. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να άρετε αυτή την αντίφαση που υπάρχει στο σημείο υπαριθμών 2 ανάμεσα στις ε, ευέλικτες ε, συμβάσεις εργασίας και τις ε, σταθερές και άκαμπτες. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να επικρατήσει μια ισορροπία. Μέχρι τώρα όλα αυτά ήταν εις βάρος των εργαζομένων. Και αν λοιπόν ε, βλέπουμε και επιτρέπουμε την αύξηση της επισφαλούς απασχόλησης και διαπιστώνουμε ότι η επισφαλής απασχόληση οδηγεί στη φτωχοποίηση, ε, αυτή, αυτό είναι το αίτιο. Το αίτιο είναι η επισφαλής απασχόληση και η ευελιξία. μας Μεζερίτσε, εκ μέρους των ε, Πρασίνων, παρακαλώ. Ευχαριστώ και εμεί θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεση. Συμφωνούμε απόλυτα με τη γενική προσέγγιση που απαιτεί δηλαδή τολμηρή αλλά και πολύ συγκεκριμένη δέσμη πολιτικών και από την Κομισιόν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο σχέδιο έκθεση υπάρχουν πολλά καλά στοιχεία, δεν θέλω να τα παριθμίσω όλα τώρα, αλλά όπω ε, λέει η εισηγήτρια ε, Πράγματι, ο κοινωνικός αυτός πυλώνας δεν πρέπει να περιορίζεται στην Ευρωζώνη, αλλά να ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ζητείται νομοθεσία σε πολλά σημεία. Παραδείγματο χάρη για το κατώτατο εισόδημα, για δίκαιε συνδικέ εργασία, οποιαδήποτε μορφή εργασία και για την κοινωνική στέγαση και τις κοινωνικές υπηρεσίες και κάτοικων βοήθεια. Επίσης, αυτό ο αργυρός κανόνα για τι κοινωνικές επενδύσει είναι κάτι πολύ σημαντικό, πρέπει να το προωθήσουμε. Και κάτι άλλο, δύο προκλήσεις και αυτά τα στοιχεία λείπουν. 60% λέει η έκθεση θα πρέπει να είναι το κατώτατο εισόδημα. Αλλά εδώ βλέπουμε διαφορέ ε, στα κράτη-μέλη λόγω ε, ε, τη διαφορετική κατάσταση. Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία. Αυτό το 60% εκεί πάλι θα άφηνα τον εργαζόμενο ε, σε κατάσταση φτώχειας. θα μπορούσαμε να θετήσουμε μία μέθοδο για τον υπολογισμό του κατώτατου εισοδήματο και θα υποβάλουμε σχετικέ τροπολογίε. Επίση, ζητείται χρηματοδότηση, επαρκή χρηματοδότηση. Όμω, για την Ευρώπη και για την Ευρωζώνη δεν αναφέρεται ότι θα πρέπει να προχωρήσει σε μια δημοσιονομική ένωση. Δεν υπάρχει, ε, και τα είδαμε αυτά, απόλυτη ολοκλήρωση στην Ευρωζώνη. Επίσης, η κοινωνική ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θα ε, μπορέσουμε να απορροφήσουμε τους κοραδασμούς και να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες και να αποφύγουμε την αναγκαστική μετανάστευση μόνο με μια στεναρή κοινωνική πολιτική. Και επαναλαμβάνω υπάρχει αυτή η δέσμευση για τη Δημοσιονομική Ένωση. Εμείς στηρίζουμε ε, το έργο της εισηγήτριας και θέλουμε απλά να συμπεριφθούν αυτά τα στοιχεία που προανέφερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι εδώ κυρία Τζέας για την ευθυντή. Η ΕΝΕΦ επίσης εκπροσωπείται εδώ. Ή ο Ντομινίκ Μάρτε. για το ΕΝΕΦ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λάρσον που ήρθε εδώ ω φερέφο του κυρίου Γιούνκερ, που δεν είναι βέβαια ακριβώς, αλλά τέλος πάντων εδώ ήρθε ω φερέφωνο και σύμβουλος του κυρίου Γιούνκερ. Πολύ ωραία έχουν αυτά στα αυτιά μας, μια ωραία μουσική που την ακούμε δεκαετίες. Και όλοι σχεδόν όσοι πήραν το λόγο ναι, είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι το μέσον ε, διαμερασμού του πλούτου, το γάλα και το ε, πρέπει να ρέουν. Ναι, πράγματι. Έγινε όμως αυτό. Τελικά διαμοιραζόμαστε, μόνο τη μιζέρια και την εξαθλίωση. Έχουμε φτωχοποίηση και το λένε όλοι τελικά. Άρα μιλάμε για μια διαπίστωση αποτυχίας, κραυγαλαία, κύριε Λάρσο. Και το ομολογείτε κι εσείς. Το Σεπτέμβριο του 2007 έγινε μια τεράστια διαβούλευση για ένα ευρωπαϊκό πυλώνα, κατόφλι ε, των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι κάτι που το υπασχόσασταν και το επαγγελώσασταν εδώ και χρόνια. Φοβούμαι. Και δεν είμαι ο μόνος που έχω ανοίξει τα μάτια μου. Το βλέπουν και πολλοί άλλοι. Αυτή η περισσότερη Ευρώπη θέλετε να επιβάλλετε σημαίνει ισοπαίδωση προς τα κάτω. Άρα ακόμη και περισσότερη μιζέρια που θα πρέπει να τη μοιραστούμε και θέλετε να μοιραστούμε όλο ο πλανήτη πλέον. Αφού πρέπει να δεχτεί η Ευρώπη 6 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ανήκουν στα πράγματα. Ένα δευτερόλεπτο μου έμεινε και θέλω να σας προειδοποιήσω. Πάτε κατευθείαν στον τοίχο να χτυπήσετε. Και ο κύριο Ζάσης σας το επενθυμίσει. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Γκυγιόν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Σύμβουλε. Εάν κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προκλήσεις, υπάρχει ο κίνδυνος ε, να καταρρεύσει κάποια στιγμή. Είναι δύσκολο να ε, ξεχωρίσουμε το κοινωνικό από το οικονομικό ζήτημα. Το είπατε και εσείς ε, προηγουμένως ότι υπάρχει το έγγραφο ακριβώς για, για την οικονομική απόκληση. Έχω δύο ερωτήματα. Πρώτον, Υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα επαρκές κοινωνικό επίπεδο στην Ευρώπη εάν παραμείνουμε ε, στη λογική της ε, απόλυτης ελεύθερης συναλλαγής με τον υπόλοιπο πλανήτη. Δεν υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ των δύο στόχων. Και ως προς αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως πρέπει να επανεξετάσει αυτή την ε, προσέγγιση των ελεύθερων συναλλαγών που βλέπουμε ότι έχει σημαντικές επιπτώσεις τις οποίες διαπιστώνουμε και σήμερα. Δεύτερον, για την εγχώρια, συγγνώμη, την εσωτερική αγορά, ε, υπάρχει όντω μια εξίσωση προ τα κάτω, αλλά ποιοι είναι οι απτοί στόχοι στους οποίου θα στηριχθείτε και τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά ε, τον ε, βασικό μισθό στο 60% του μέσου μισθού, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Γιούτε Στάινμπρουκ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τόσο από Εγώ πιστεύω ότι όταν υπάρχει συνεργασία στην Ευρώπη μπορούμε να λύσουμε προβλήματα. Σχετικά με την ανεργία, μπορούμε αυτό να το εξηγήσουμε στους πολίτες. Ε, αυτή την εισαγωγή ήθελα να κάνω και θέλω τώρα να κάνω τις ερωτήσεις μου. Ο Jean-Claude Juncker ε, υποσχέθηκε το τριπλό αλφα για την κοινωνική Ευρώπη. Και εγώ το βρίσκω πάρα πολύ καλό που δουλεύουμε πάνω στον κοινωνικό πυλώνα, γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται ε, συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Και ερωτώ ε, τον κοινωνικό πυλώνα πώς πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε ως στήλο, ως σημείο αναφοράς, ως συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις ε, οι οποίες χρειάζονται ορισμούς ε, για τις ε, κοινωνικούς καταλόγους, τις κοινωνικές προδιαγραφές. Αυτό το είχε υποσχεθεί ο κύριος Γιούγκερ. Χρειαζόμαστε μια αγορά εργασίας η οποία να ε, χρειάζεται κοινέ ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό θα προκύψει σχετικά γρήγορα. Γιατί ξέρετε, εμένα στη δική μου την εκλογική περιφέρεια εξακολουθούν να με ρωτάνε τι έγινε, και τι θα γίνει με την υπόσχεση του κύριου Γιούγκερ η υπόσχεση του κύριου Γιούγκερ θα υλοποιηθεί σε αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να και τον κύριο Λάρισον και δύο έχουν δίκιο. Και η συγγήτρια αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σήμερα να έχουμε μια καλή συζήτηση και πιστεύω ότι το περιεχόμενο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον διότι εμείς επιθυμούμε να επιτύχουμε κάτι για πάρα πολλούς ανθρώπους όχι μόνο για μας τους λίγους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμούμε περισσότεροι άνθρωποι ε, να μπορούν να έχουν μια καλή και λογική απασχόληση. Εδώ λοιπόν στην Επιτροπή Απασχόλησης έχει κανεί συχνά την εντύπωση ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από τους ανθρώπους και από τα καθημερινά τους ε, προβλήματα. Μιλάμε συχνά για το μέλλον και νομίζω ότι και σε αυτή την έκθεση βέβαια γίνεται λόγος για το μέλλον. Ελπίζω όμως ε, πρώτα απ' όλα αυτό που θα ενδιαφέρει είναι να αναζητήσουμε την επαφή με τους ανθρώπους ε, έξω από του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν είχαμε αυτή την ε, επαφή, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε πάρα πολλά και θα καταλήγαμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για ε, τον κοινωνικό πυλώνα, αλλά μέσα στις συνθήκες θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος κοινωνικού πρωτοκόλλου. Και νομίζω ότι τώρα πια υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εγώ όλα αυτά εδώ τα βλέπω ως το βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μέχρι τώρα αγωνιστήκαμε ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Κοινοβούλιο για να υπάρχει μια κοινωνική ατζέντα, μια διαφορετική Ευρώπη. Αν όμως μπορούμε να τα θεμελιώσουμε όλα αυτά στι συνθήκε, τότε παίζουν και ένα ρόλο και θα λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη. Ελπίζω λοιπόν ότι ο κύριος Λάρσον, η Μαρία Ζωάου και όλοι οι άλλοι ε, σε αυτήν την Επιτροπή θα συνεχίσουν τις εργασίες ε, προς αυτή την κατεύθυνση γιατί πιστεύω ότι ε, χρειαζόμαστε ευρεία υποστήριξη για να τα πετύχουμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πυρίνσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό ε, με την αξιολόγηση αυτής της έκθεσης, ότι δηλαδή προωθεί σημαντικά την έννοια του κοινωνικού πυλώνα. Θεωρώ ότι πραγματικά ε, ε, έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα σε σχέση με τι προηγούμενε προτάσει τη Επιτροπή. Ανέφερε ο κ. Λάρσεν ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν φιλικά ούτε προ τι επιχειρήσει ούτε προ του εργαζόμενου. Όπω αναφέρεται και στο επεξηγηματικό σημείωμα, ε, ήταν εξαιρετικά φιλικό όμως αυτό το διάστημα προς τις τράπεζες, γιατί σχεδόν 2-3 ευρώ ε, των χρημάτων των φορολογουμένων δόθηκε εν είδη κρατικής επιχορήγησης ε, στον τραπεζικό κλάδο από το 2008 μέχρι το 2014. Και τώρα έχουμε ένα τεράστιο επενδυτικό κενό και όλα αυτά τα μέτρα λιτότητας που πλήττουν κατά κύριο λόγο τις κοινωνικές δαπάνες. Αναφερθήκατε σε αυτό που λένε ο κύριος Δράγκη, η κυρία Λαγκάρτ και τα όσα αναφέρθηκαν ε, εκτός ε, ε, τη συζήτηση, στο περιθώριο της συζήτησης ε, στο G20 είναι ότι χρειαζόμαστε μια αλλαγή παραδείγματος και αυτή η αλλαγή σε τελική ανάλυση θα πρέπει να μας οδηγήσει όχι μόνο σε μια οικονομική και νομισματική ένωση, αλλά σε μια οικονομική, κοινωνική και νομισματική ένωση. Όπως ε, αναφέρθηκε το να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να έχουμε ανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική διάσταση και τη διαμόρφωση κοινωνικής εταιρικής σχέσης που παράγει πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη. Έχω λοιπόν τα εξή ερωτήματα. Εισάγεται προτάσεις για αυτή την αλλαγή, σε μια αντίστοιχη αλλαγή ισοδύναμη στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και πώς θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει νομική εφαρμογή και υλοποίηση των όσων συζητούμε. Ευχαριστώ. Ελίζα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο Ροντρίγκε ε, για την ενασχόλησή της ε, με αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά φλέγον το ζήτημα σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ε, το σύνολο των, Ευρωπαϊκών, των Ευρωπαίων πολιτών θα ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στην Ευρώπη μόνο εάν εμείς είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε αυτό τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Και είμαι απόλυτα πεπισμένη αυτό το που σας λέω. Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερως δύο σχόλια, δύο ερωτήσεις που θέσατε. Πρώτον, η απόκληση μεταξύ της αγοράς απασχόλησης και του συστήματος επανεισαγωγής στην αγορά επασχόλησης. Πώς μπορείτε να μας διευκρινίσετε περαιτέρω αυτή την απόκληση. Τα 10 επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη απασχολησιμότητα σήμερα δεν υπήρχαν πριν από 10 χρόνια. Το διοικητικό σύστημα επανεισαγωγής στην αγορά εργασίας ε, αδυνατεί δηλαδή να ακολουθήσει την ταχύτητα ε, της ε, εξέλιξης των επαγγελμάτων. Ποιο είναι το πρόβλημα ακριβώ εδώ ποια είναι η δυσκολία να επανεσαχθούν και να επανανταχθούν μάλλον οι συμπολίτε μας στην αγορά απασχόληση. Το δεύτερο, είπατε ότι δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε πλέον στις ε, καταρτήσεις, αλλά στις δεξιότητες και τις ικανότητες. Εγώ εδώ καιρό είμαι κάθετα πεπισμένη ότι εάν δεν αναπτύξουμε την επανένταξη στην αγορά απασχόλησης μέσω της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, και από την επαγγελματική σταδιοδρομία αλλά και από την αρχική εκπαίδευση δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα γιατί υπάρχει μια τεράστια ταχύτητα εξέλιξης, ανάπτυξης ε, και εξέλιξης των επαγγελμάτων που δεν ε, αντιστοιχεί στον ρυθμό εξέλιξης της, επαγγελ... της εκπαίδευσης μάλλον. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε πρότυπα λοιπόν από κάτι που είναι πολύ πιο ε, λειτουργικό για το σύνολο των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπροκ παρακαλώ.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 αυτή τη συζήτηση πάρα πολύ καλή τη βρήκα και κυρίως αυτά που μας είπε και ο εκπρόσωπος του κυρίου Γίνκερ γιατί είχαμε τη δυνατότητα ε, να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις ε, διαφωνίες που υπήρχαν δηλαδή ότι δίθεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην υποθέμενη ε, δημοσιονομική σοβαρότητα αφενός και αφετέρου στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για την οικονομική πολιτική και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι η κοινωνική πολιτική έχει νόημα ε, μόνο εφόσον ε, συζητείται και μπορεί να παίξει ρόλο σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη και την ε, ε, το δημοσιονομικό μοντέλο και με την κοινωνική ειρήνη, γιατί και αυτό είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Αυτό φαίνεται ότι δεν το γνωρίζουν, δεν το έχουν ε, κατά νου όλοι οι εργοδότες. Αυτό είναι λάθος, νοηματικό λάθος. Πιστεύω λοιπόν ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι συνθήκες κάτι μπορούμε να κάνουμε. Τα επόμενα 8 χρόνια δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τροποποίηση των συνθήκων και λόγω του ότι υπάρχουν και συγκεκριμένε προϋποθέσεις για διακοινωνία κυβερνητικέ, για διαδικασίε κυρώσεων. Αυτά είναι όνειρο θερινή νυχτό. Το, το είχα και εγώ παλιά το όνειρο αυτό, αλλά δεν πρέπει να θεωρούμε ότι σήμερα μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι μπορεί να επιτύχουμε ε, τροποποίηση των συνθήκων ακόμα και αν το επιθυμούμε διακώς, ακόμα και αν θέλουμε να υπάρξουν τροποποίηση των συνθήκων. Ξέρετε, μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι πολλοί επικαλούνται αυτό το, την τροποποίηση ως άλλοτη για να μην κάνουν τίποτα στην πρακτική. Και ε, βλέποντας την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, αν τη θυμάμαι καλά, νομίζω ότι ε, το θέμα, ε, το κοινωνικό, όπως και το θέμα του περιβάλλοντος είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Θα εκμεταλλευτούμε λοιπόν τις δυνατότητες που υπάρχουν. Αυτό νομίζω ότι αξίζει να το ερευνήσουμε και κατά πόσο θα το κάνουμε στο Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν ή το κατά πόσο θα το κάνει ο νομοθέτης. Δηλαδή επισημένοντας ε, το ότι ε, πρέπει να γίνεται αναφορά στις συνθήκες. Ε, νομίζω ότι έτσι μπορούμε να προάγουμε λιγάκι το ε, μοντέλο της απασχόλησης. Ο κύριος Φουντούλης παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Γιούγκερ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα ευχολόγιο που απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται οι κοινωνικές ανισότητες στην Ευρώπη να είναι τόσο μεγάλες Μα οι ίδιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν σε ανισότητες στην Ένωση και στην ανεργία και στη φτώχεια. Η Ευρώπη γερνάει, όπως λένε όλοι. Αλλά δεν είδαμε να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της οικογένειας και να δώσει κίνητρα για να γεννιούνται νέοι Ευρωπαίοι. Αντίθετα, έχουμε καλέσει στην Ευρώπη όλους τους οικονομικούς μετανάστες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φτηνά εργατικά χέρια για τις βιομηχανίες. Οι ευέλικτε μορφέ απασχόληση έχουν δώσει το δικαίωμα στι μεγάλε εταιρείε να κερδοσκοπούν ει βάρο των εργαζομένων και οι εργαζόμενοι να ζουν στο όριο τη φτώχεια και να πληρώνονται λιγότερε ασφαλιστικέ εισφορέ, τα οποία με σκοπό έχουν να διαλύσουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Με τι πολιτικέ των μνημονίων και των μέτρων λιτότητα που επιβάλλονται στι οικονομικά ασθενέστερε χώρε, ένα είναι σίγουρο. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν εξακολουθεί να αγκαλιάζει τόσο σφιχτά τι χώρε αυτέ, με αποτέλεσμα να του δημιουργεί ασφυξία, κάποια στιγμή θα αποφασίσουν να απεγκλωβιστούν από αυτή την αγκαλιά. Ευχαριστώ. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, temos as maiores reservas quanto eh, Ευχαριστώ. Σε σχέση με τον πυλώνα αυτό έχουμε κάποια ζητήματα. Ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, η οικονομική και η χρηματοπιστωτική κρίση, γίνεται λόγο εδώ για κάποιου κοινωνικού δείκτες, για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. και είναι κατά των εθνικών ε, συμφερόντων ε, των εργαζομένων. Αυτή ε, την πορεία μόνο τα μεγάλα κεφάλαια και οι πολυεθνικές θα ωφεληθούν. Μεγάλη κρίση βιώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πυλώνας αυτός είναι σαν να, θέλουμε να συγκαλύψουμε ε, με κάποια, με ένα μικρό μακιγιάζ την οικονομική διακυβέρνηση που είναι το κύριο στοιχείο. Και βλέπουμε και στην πράξη ότι ούτε οι στόχοι επιτυγχάνονται παρά μόνο οι συσσόρες της οικονομικής εξουσίας. Πώς συμβαδίζει αυτό το καπιταλιστικό project που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κοινωνικά δικαιώματα. Τελικά προωθείται η εργασιακή μεταρρύθμιση που θα οδηγήσει σε εναρμόνιση. Και όλα αυτά υπέρ της εργοδοσίας. Σας ανησυχεί το έλλειμμα. Μην πάτε ενάντια όμως στους εργαζομένους υπάρχει το κοινωνικό, κοινωνική σύμβαση. Στην Πορτογαλία καταστρέφονται. Μειώνονται, πέφτουν στο κενό προσπάθειες, οι μισθοί, κατώτατοι μισθοί έχουν στην Πορτογαλία σοπεδωθεί. Μην παρεμβαίνετε λοιπόν στις εθνικές κοινωνικές πολιτικές των κρατών με εκβιασμό και με κυρώσεις όπως αυτές ε, που υπέστη η Πορτογαλία. Μην επιτίθεστε στα εργασιακά δικαιώματα αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, ο κοινωνικός πυλώνας δεν θα είναι επίτευγμα, αλλά θα συνεχίσει να επιτίθεται κατά των δικαιωμάτων των εργαζομένων, θα αυτοδηγεί σε φτωχοποίηση και κοινωνική εκμετάλλευση. Τελευταίο ομιλητή Μόρτεν Λόκεγκαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Λάρσον. Ήταν ενδιαφέρουσα η παρουσίαση περισσότεροι εξημών συμφωνούμε νομίζω με τον κύριο Γιούγκερ ότι χρειαζόμαστε μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Αλλά υπάρχει και ένα ερώτημα ίσως πιο ουσιώδες. Πώς θα την πετύχουμε αυτή την κοινωνική Ευρώπη. Και αν συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική θα πούμε κοινωνική Ευρώπη περισσότερη σημαίνει πως και μια κοινωνική ένωση. Συμφωνώ με τους συναδέλφους ε, ότι χρειάζεται ε, αυτή η συζήτηση σε ένα πιο ευρύτερο ακροατήριο, ένα πιο ευρύτερο κοινό. Γι' αυτό και θα αλλάξω γλώσσα τώρα και θα μιλήσω από εδώ και πέρα στα δανέζικα. Όπως έλεγα λοιπόν κύριε Λάρσον, έχω μια ερώτηση σε σχέση με την παρουσίασή σας. Διότι αν εξετάσουμε την κατανομή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, λέμε για την ευελιξία με ασφάλεια, το λεγόμενο flex security, αλλά για τροποποίηση των συνθήκων δεν γίνεται λόγος ουσιαστικά. Δεν είναι ότι μας ενδιαφέρει βέβαια και τόσο πολύ κάτι τέτοιο, αλλά... Κύριε Λάρσον, υπ' αυτή την ε, οπτική γωνία έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας κάτι τέτοιο, μια τροποποίηση συνθήκων. Σε ό,τι αφορά το flexicurity, ε, πολλοί έχουν κρουστόν τον ε, κόδωνα του κινδύνου 4,2 είναι η ανεργία στη Δανία. Που σημαίνει ότι όσο πιο ευέλικτη είναι μια αγορά εργασία, τόσο περισσότερε θέσει εργασία υπάρχουν. Μπορείτε να μα το επιβεβαιώσετε ότι βλέπετε και εσεί τα πράγματα. Λοιπόν, πολλά τα ερωτήματα προς τον ε, κύριο Λάρσον. Ε, θα ήθελα να του δώσω τέσσερα λεπτά, ε, μετά στη Μαρία Ζωάου ένα λεπτό για να κλείσει το θέμα γιατί νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει λιγάκι. Παρακαλώ. Ε, θα είμαι σύντομος. Άκουσα τις απόψεις σας και τα σχόλιά σας ε, και αυτά που είπατε. Τα έβρικα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και μοιάζουν πάρα πολύ με όλα αυτά που ακούω και στα κρατη θα συμπεριλάβω τα σχόλιά σας ε, στις συζητήσεις που θα κάνουμε. Θέλω να τοποθετηθώ μόνο σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Και αυτό ε, διότι δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που θέσατε. Ε, πρώτα πρέπει να γίνουν διαβουλευσει ε, και μετά να προκύψουν απαντήσει. Δεν μπορεί όταν εγώ είμαι εδώ να ε, γίνουν, να δοθούν οι απαντήσεις. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Μία συγκεκριμένη ερώτηση είναι η εξή. Θα υπάρξουν περισσότερες προτάσεις. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Αυτό δεν είναι ένα έγγραφο που να είναι όλα προμαγειρεμένα. Ε, μαγειρεύονται. Τώρα ε, θα αποκτήσει περιεχόμενο, μεγαλύτερο περιεχόμενο το έγγραφο. Γι' αυτό λοιπόν η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ναι. Το πώς βέβαια θα γίνουν όλα αυτά θα το δούμε. Θα τα δούμε στις αρχές του επόμενου έτους όταν θα εξαχθούν τα συμπεράσματα. Νομίζω δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω και προσφέρω και το χρόνο μου στους ε, υπόλοιπους μιλητές. Ε, είσαστε ένας καταπληκτικός επαγγελματίας ε, και ένας ευγενής κύριος παλαιάς κοπής. Η Μαρία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό που είχαμε μια τόσο πλούσια συζήτηση με έγκυλο ενδιαφέρον πολλών μελών της Επιτροπής, αλλά και του κυρίου Λάρσεν. Τον γνωρίζω πολύ καλά και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται εδώ μαζί μας με την ιδιότητα του Συμβούλου του Πρόεδρου Γιούνκερ. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο οφείλει να οργανώνει τις εργασίες του με κατάλληλο χρονικό πλαίσιο για να είναι έτοιμη η έκθεση πριν προετοιμάσει το Σώμα των Επιτρόπων ε, την πρότασή του. Και νομίζω το χρονοδιάγραμμά μας είναι καλό προς αυτόν τον σκοπό. Μπορούμε να αποφεληθούμε τις δημόσιες διαφούλευσεις που λαμβάνει η χώρα και συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να ανοίξουμε το Κοινοβούλιο προς τους Ευρωπαίους πολίτες και την Ευρωπαϊκή Εάν ολοκληρωθεί η έκθεση μέχρι τον Ιανουάριο, νομίζω ότι εντάσσεται πολύ καλά στο χρονοδιάγραμμα τη Επιτροπή. Δεύτερον, καλούμαστε να δώσουμε επικαιροποιημένε απαντήσει σε νέε προκλήσει. Ήθελα μόνο να επισημάνω ότι ναι, πρέπει πολύ καλύτερα να οργανώσουμε τη συμπερίληψη των νέων ε, και των γυναικών και την ένταξή του ε, στην αγορά εργασία. είναι, αυτά είναι δύο ζητήματα που πρέπει να τα πάμε πολύ καλύτερα. Δεύτερον, οι επιπτώσει της ψηφιακή επανάστασης. Πρόκειται για νέες μορφές απασχόλησης που θα ανοίξουν ευκαιρίες, όμως πρέπει να διασφαλίσουμε την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τέλος, για τα μέσα για να έχουμε μια αξιόπιστη έκθεση θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι για τους στόχους, τα μέτρα και τα μέσα που θα επιστρατεύσουμε, τα οποία είναι νομοθετικά, αλλά και μέσα διακυβέρνησης. Πρέπει καλύτερα να συντονίζουμε τις ε, οικονομικές και και κοινωνικέ πολιτικέ. Και τρίτον, χρηματοδότηση, οικονομική πόρη. Γιατί εάν έχουμε κατά νου τεράστιε κοινωνικέ επενδύσει, θα πρέπει να έχουμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα στον κοινωνικό πυλώνα. Θα πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα απτά μέσα. Επομένω, ε, βασίζομαι στους συναδέλφους να είναι αρκετά τολμηροί και με τη σειρά μας να καλέσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστούμε πολύ Μαρία. Επιτρέψτε μου να κάνω κι εγώ μία παρατήρηση ε, πριν τελειώσουμε. Δηλαδή, ξέρετε, εγώ δεν πήρα μέχρι τώρα το λόγο, γιατί, ξέρετε, άκουσα έτσι χαμογελώντας μόνος μου ότι πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες. Ξέρετε, κι εγώ έτσι το βλέπω. Όμως δεν έχουμε ούτε τις πολιτικές συνθήκες, ούτε το χρόνο να επιτύχουμε κάτι τέτοιο κατά τα επόμενα έτη. Παρόλα αυτά όμως ε, θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο, διότι η κοινωνική ρήτρα πρόοδου στις ε, συνθήκες ε, λείπει από τις συνθήκες σαν να είναι ένα γονιδιακό ελάττωμα. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της τροποποίησης των συνθήκων και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Δηλαδή μια αδικαιολόγητη συμπεριφορά, δημιουργείται ένας ενδιάμεσος χώρος και αυτό έχει τον τίτλο νομοθετικά μέτρα τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω λοιπόν να σας υπογραμμίσω αυτό που έχω πει και παλαιότερα. Για αντισυμβατικές αλλαγές, αυτό δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει. Δεν χρειάζονται οι άνθρωποι κάτι τέτοιο, θα συμβεί το αντίθετο. Γι' αυτό λοιπόν ε, σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, πρέπει να υπογραμμίζεται ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προχωρήσει η κοινωνική Ευρώπη. Αυτά είχα να σας πω εγώ με τις ε, θερμότερες ευχές μου προς τον κύριο Γιούγκα. σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λάρσεν και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. So. Yes, friends, then we proceed to... Αγαπητοί φίλοι, να περάσουμε στο σημείο 8 της ημέρησιας διάταξης. Δηλαδή την ανάγκη για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τον τερματισμό και την πρόληψη του χάσματος ε, στη συντάξη ανάλογα με το φίλο. Η κυρία Γκονθάλεφ Πένιας έχει το λόγο. Δύο λεπτά για την εισαγωγή. Ευχαριστώ. Νόμιζα ότι είχα πέντε λεπτά στη διάθεσή μου για να σας παρουσιάσω το σχέδιο νομοδότησης Η πρόεδρος. Δυστυχώ χρειάστηκε να προσαρμοστούμε γιατί θα έχουμε και την ψηφοφορία σε λίγο. Δυστυχώ δεν μπορώ να σα δώσω πάνω από δύο λεπτά. Μάλιστα. Θα προσπαθώ να τα πω πιο γρήγορα. Ε, και θα σας παρουσιάσω λοιπόν το προσχέδιο της γνωμοδότησης στην ανάγκη μιας στρατηγικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το ερματισμό και την πρόληψη της, του συνταξιδοτικού χάσματος ανάλογα με το φύλλο. Είχα δέκα βασικά επιχειρήματα για να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες και τα στοιχεία που δημιουργούν αυτό το χάσμα σε ό,τι αφορά την ποσότητα, τη διάρκεια και τις συνθήκες ε, των ε, συντάξεων. Και ήθελα να προτείνω και κάποια μέτρα για τη διόρθωση αυτού του χάσματος. Πρώτον, ε, το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη είναι απαράβατο και σίγουρα θα πρέπει να μην παρεμβάζεται και το θεμελιώδες δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο δεν γίνεται σεβαστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης όρις η ισότητα ανακοινών αναγνωρίζεται από πολλές συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, το αναγνωρίζουν και πολλά τα συντάγματα των κρατών μελών για αξιοπρεπείς δημόσιες συντάξεις, δηλαδή, χωρίς διακρίσεις και στο πλαίσιο εξωτικών συστημάτων που θα είναι οικουμενικά υποχρεωτικά αλληλέγγυα, επαρκή, αναδιανεμητικά βιώσιμα. Για όλους αυτούς τους λόγους Ευθύνη μας είναι να διορθώσουμε τις δυσκολίες αυτές. Γι' αυτό και προτείνουμε κάποια μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη, κατώτατη, εγκυμένη κατώτατη σύνταξη για όλα τα άτομα άνω των 65, ενίσχυση των συνταξιδοτικών συστημάτων, με εισφορές φορολογικά πρόδευ... με αύξηση προοδευτική κλίμακα, συμπέριψη μηχανισμών για να μην επηρεάζει αρνητικά ε, η φροντίδα κάποιου ηλικιωμένου κάποιου παιδιού και επίσης ε, μερική απασχόληση και έπλης απασχόληση, να μην έχουμε διακρίσεις στις συντάξεις λόγω των ήδη φυστάμενων διακρίσεων στο πλαίσιο ε, της αμοιβόμενης εργασίας και της ε, ε, κατοίκων φροντίδας και συμφιλίως επαγγελματικού γενιακού προσωπικού βίου και ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε μια δίκαιη αγορά εργασία, περισσότερη δημόσια χρηματοδότηση για βελτίωση των υποδομών, δωρεάν υποδομών, για παροχή ε, σε ηλικιωμένου και παιδιά. Κατώτατο μισθό, 60% του μέσου μισθού και επίσης πολιτικές λιτότητας και ό,τι ε, μέτρο βασίζεται στη δημοσιονομική βιωσιμότητα να μην πλήττουν ε, τη συντάξη, αξιοπρεπή συντάξη ιδίως των γυναικών. Ελπίζω να εργαστούμε με υπευθυνότητα και περιμένω τα σχόλια και τις τροπολογίες σας. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Κυρία Κοσλόσκα είναι εδώ. Όχι. Σου πει κάποιο άλλο το ΕΛΚ. Παρακαλώ κύριε Σεντέρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι εδώ κυρία Κοσλόφσκα, επομένω θα ήθελα να αναγνώσω τα σχόλια που έχει προετοιμάσει. Το συντεκτικό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι βασικός δείκτης για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων εν γέννη, γιατί αντικατοπτρίζει τα μειονεκτήματα τα οποία βιώνει η γυναίκα καθ' όλη τη διάρκεια της ε, σταδιοδρομίας της. Το στεξιωτικό χάσμα μεταξύ φύλων δεν τεκμηριώνεται και εξηγείται μόνο από τις διακρίσεις και από τα στεξιωτικά συστήματα, αλλά προκύπτει και από την άνηση θέση της γυναίκας στην απασχόληση, που χαρακτηρίζεται από τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον, χαμηλότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Δεύτερον, όταν η γυναίκα είναι ανεργή τότε ε, τίνει να επιλέγει δουλειές που, ε, με, χαμηλό, ώρες και κατά μέσο ώρα, όρο οι γυναίκες ε, αμείβονται με χαμηλότερους μισθούς. Για αυτούς τους λόγους πλέον αποτελεσματική και οικονομικά αποθετική λύση μακροπρόθεσμα για την μείωση του συνδεκτικού χάσματος μεταξύ των φύλων είναι να διασφαλίσουμε μια ισότιμη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. με πολιτικές που έχουν ως σκοπό τη συμφιλίωση του επαγγελματικού και προσωπικού βίου. Αυτή η θέση θα αντικατοπτριστεί αντικατοπτριστεί και στι ε, τροπολογίε που θα υποβάλει η κυρία Κοσλόφσκα εξ ονόματο του ΕΛΚ ε, προκειμένου να ε, διασφαλίσουμε ότι θα τηρείται η αρχή της επικουρικότητας. Είναι σημαντικό η γνωμοδότηση αυτή να συνάδει και με τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Στάινρουκ από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κυρία Μπλίνκεβιτσούτε. Δυστυχώ σήμερα δεν μπόρεσε να έρθει. Η Σκέωδη Συγκήτρια ευχαριστεί για μια πολύ καλά προετοιμασμένη γνωμοδότηση με πολλέ ιδέε και εκ μέρου των σοσιαλδημοκρατών. Λείπουν κάποια σημαντικά θέματα τα οποία εμεί θα τα συμπληρώσουμε. Εμά μα ενδιαφέρει η κρατική σύνταξη, δηλαδή η Συγκήτρια υπογραμμίζει τη σημασία τη κρατική σύνταξη. Μα ενδιαφέρει όμω και ε, το δεύτερο δεύτερο σκέλος του πυλώνα, η ε, επιχειρησιακή, η επικουρική σύνταξη αν θέλετε, επικουρικές λοιπόν, το τι ε, αποφασίζεται μετά από συλλογικές διαπραγματεύσεις και να υπάρχει και ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Η ιδιωτική σύνταξη ε, και δυνατότητα σύναψη συνταξιωτικού ιδιωτικού συμβολέου, αυτό δεν πρέπει που δεν είναι να το σκεφτούμε. Γιατί αυτό αφορά μόνο εκείνου ε, που είναι πλούσιοι. Γι' αυτό λοιπόν εμείς προβλέπουμε για τα κράτη-μέλη σε περίπτωση συνταξιωτικής μεταρρύθμισης να τα λάβουν όλα αυτά υπόψη και επιπλέον επιθυμούμε να καταβληθούν και περαιτέρω προσπάθειες ε, για να υπάρξει πρόοδος που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε απόλυτη διαφάνεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος, ε, εκ μέρους της ΙΣΙΑΡ Γιάννα Τσιτάνσκα. Ευχαριστώ. Συζητούμε τα συνταξιδοτικά συστήματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τονίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει παρά περιορισμένα δικαιώματα στον τομέα αυτό. Εμεί ουσιαστικά είμαστε ένα φόρμα ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ακόμη και όταν είναι καλοπροαίρετε οι προτάσει να σεβόμαστε τι διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών. Επίση υπάρχουν πολύ άγνωστοι ε, χ, πολλέ άγνωστε παράμετροι. Βελτιώνεται σίγουρα το εισόδημα των γυναικών σε πολλέ χώρε, αλλά δυστυχώ σε ό,τι αφορά τι συντάξει βλέπουμε να μην αντικατοπτρίζεται αυτό. Οι συντάξει επηρεάζονται από διάφορου παράγοντε και πολύ δύσκολα μπορούμε να μετρήσουμε σε αυτού του παράγοντε, όπω είναι η λήψη ποιοτικών δεδομένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να υπολογιστούν αυτέ οι διαφορέ ε, όλα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια προσθέμενη εξή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να ασκήσουμε πιέσει ε, για να μπορούν να λαμβάνονται πιο τεκμηρωμένε αποφάσει. Δεύτερον, οι γυναίκε που φροντίζουν είτε εξαρτημένα άτομα είτε ε, παιδιά είναι ευάλωτε όταν μεγαλώσουν ηλικιακά, γιατί υπάρχουν μεγάλα κενά στη σταδιοδρομία του και αυτά αντικατοπτρίζονται και στη σύνταξη που θα πάρουν στο τέλο και στο, στο βιωτικό επίπεδο που θα έχουν όταν συνταξιοδοτηθούν. Εκεί πρέπει να σχέσουμε πίεση τα κράτη-μέλη, να αντισταθμίσουν τα κενά αυτά στην ε, ενεργό ε, φάση της ζωής μιας γυναίκας για να, μπορεί, να έχει και μια εξωπρεπή σύνταξη. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλά πάει το 1,5 λεπτό κάθε Να το κάνουμε και στο μέλλον. Για να τον επόμενο συμμιλητής δεν είναι εδώ. Τερέρα, εκ μέρου των Πρασίνων, δεν βλέπω να υπάρχει. Εκ μέρους των Πρασίνων, παρακαλώ, εσείς έχετε τε λόγο. Εγώ εκπροσωπώ τη Σκιώδη, η Σιγήτα Τερεράν και που δεν μπορούσε να εδώ σήμερα. Θέλω να συγχαρούμε τα την εισηγήτρια. Συμφωνούμε με αρκετές από τις υποδείξεις και προτάσεις της. Και εκτιμούμε όλους ιδιαίτερως και το ότι διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις. Θέλω να τονίσουμε που είναι πολύ σημαντικό η γυναίκα να έχει μια επαρκή σύνταξη και θα καταθέσουμε τροπολογίες για να διατυπώσουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά. Για παράδειγμα, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ευρωπαϊκά πρότυπα για το λεγόμενο care crediting ε, στα συνταξιδοτικά συστήματα. Να παίρνουν πόντους δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες φροντίζουν ηλικιωμένο ή ένα παιδί. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν πάντο δυνατόν ώστε να βοηθούν με ένδικα μέσα ε, σε περίπτωση χωρισμού ή διαζυγίου, ώστε η γυναίκα να έχει επαρκή ε, σύνταξη επίσης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα καταθέσουμε υπομορφή συγκεκριμένων τροπολογιών. Ευχαριστώ. Η Λάουρα Ατζέα δεν είναι εδώ. Ζωάν Μιλά. Κύριος Μαρτάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερα ευρύ το ζήτημα και είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς με την κυρία Συγήτρια για τις ε, προτάσεις που κάνει υπό αυτή την έννοια. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά. Πού θα βρείτε τα χρήματα. Ήδη σε πολλά κρατημέλη, κυρίως στη Γαλλία, μας λένε ότι μας τελείωσε το συνταξιδοτικό σύστημα όπως το ξέρουμε σήμερα. Δύο λύσεις που έχουμε είναι η επιμήκυνση του εργάσιμου βίου, 62, 65, κάποια στιγμή και 70 χρόνια θα αργήσει και αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται αυξάνεται το προσδόκιμο ζωή. Ε. Βέβαια, στη Γαλλία τον τελευταίο χρόνο έχει αναστραφεί αυτή η τάση από ό,τι βλέπουμε. Στατιστικά στοιχεία αυτό δείχνουν. Και δεύτερον, έχουμε την δεύτερη λύση, την μείωση και περικοπή των συντάξεων. Βέβαια, πολύ καλά τα όσα μα παρουσιάζεται. Όμω, λέτε ότι είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα, το ζήτημα αυτό, γιατί υπάρχει τεράστια ανισότητα μεταξύ κρατών μελών. Σε κάποια κράτη-μέλη ε, σχεδόν δεν υπάρχουν συντάξει και βεβαίω υπάρχουν και τα ζητήματα των ε, δύο φύλων. Προκύπτει από τις ε, εργασίες, θέσει εργασία, τις οποίες καλύπτουν συνήθως ε, οι γυναίκε. Συμφωνώ λοιπόν με όλα αυτά που είπατε, αλλά πώ με ποια χρήματα, ποιο το αναλάβει ε, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια πανευρωπαϊκή στρατηγική για να αποφεύγονται διαφορετικέ συντάξει. Ακόμα και αν στο τέλο τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που πρέπει να εφαρμόσουν τέτοιο πρόγραμμα. Όμω πρέπει να πετύχουμε το εξή. Να βρούμε στοιχεία. Στην πόλη Γερμανία ε, μας απασχολεί αυτό, ε, πού ακριβώς υπάρχουν διαφορές, κυρίως στις μητέρες. Οι γυναίκες ε, δεν υπολογίζεται στις ε, γυναίκες η εκπαίδευσή τους. Λέμε ότι θα πρέπει οι γυναίκες να βγουν στην αγορά εργασίας. Μα το θέλουν, το θέλουν οι σύζυγοι τους. Έχει κανείς σκεφτεί ότι θέλει κανείς να είναι απλώς μητέρα ή πατέρας χωρίς να πρέπει να εργάζεται. Έχετε σκεφτεί ότι μία μητέρα με τρία παιδιά δεν έχει άλλη επιλογή. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για τις συντάξεις θα πρέπει να μιλήσουμε και με τις ίδιες τις γυναίκες. Συμφωνώ με τον συνάδελφο, ε, θα πρέπει ε, να υπολογίζεται και ο χρόνος εκπαίδευσης που καταναλώνουν οι γυναίκες. Ε, υπόθηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα εγγυημένο εισόδημα όπως και στις συντάξεις το λέμε αυτό, αλλά ε, εγώ πιστεύω ότι Εάν υπολογίσουμε την εκπαίδευση των γυναικών, αυτό θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό από το να γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το χάσμα γενναιών που δεν είναι και ακριβώς σαφές τι εννοούμε. Thank you, thank you very much, um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα αυτό, το χάσμα του εξοδοτικού μεταξύ των δύο φύλων. Εμείς όμως ως Κοινοβούλιο, ε, σε ποια θέση βρισκόμαστε δεν είναι εθνική αρμοδιότητα αυτά τα θέματα. Και είναι ένα άκρος πολύπλοκο τοπίο αυτό του ε, το, το συνταξιοδοτικού. Εμείς έχουμε πρώτο πυλώνα, δεύτερο πυλώνα στη Δανία, άλλοι ε, έχουν άλλες λύσεις, ίσως ενιαίες. Επομένως, ακόμα χειρότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να λάβουμε ε, μια ομοιόμορφη να προωθήσουμε μια ομοιόμορφη λύση που δεν υπάρχει σε επίπεδο κρατών μελών. Αύξηση κατώτα των μισθών, ε, φορολογικές συμβάσεις, ε, ε, ελάχιστο αριθμό χρόνων εισφορά κτλ. Όλα αυτά είναι εκτό των αρμοδιότητων της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ενδιαφέρουσα είναι αυτή η συζήτηση, όμως τα κράτη-μέλη είναι αυτά που πρέπει να συζητήσουν, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να μάθουν το ένα από το άλλο. Οι νομοθετικές προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε, ε, από τη στιγμή που δεν έχουμε καμιά αρμοδιότητα, δεν είναι και καλύτερη λύση. Ευχαριστούμε πολύ. Απλά στον τελευταίο μελητή να του πω ότι ήδη κατά την προηγούμενη θητεία ε, μας ε, απασχόλησε το θέμα αυτό. Ε, ασχοληθήκαμε με λευκές και πράσινες βιβλούς για παράταση του χρόνου εργασίας οι αρμοδιότητες λοιπόν αυτού του Κοινοβουλίου, όσο, λι, όσο περισμένες και αν είναι για θέματα συνταξιοδότησης, ε, δεν μπορούμε να τις απορρίπτουμε όταν δεν μας αρέσει κάτι. Ε, σε άλλα θέματα η Κομισιόν ήταν πολύ πιο πρόθυμη και ε, είπε ότι ναι, αυτά τα θέματα θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα λέω όλα αυτά γιατί ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε καταρχήν επ' αυτών για να ξέρουμε πώς θα εργαστούμε. Πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Εμίλιαν Πάβελ, έκθεση εφαρμογής σχετικά με το Erasmus. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μου φτάσουν τα λεπτά που μου δώσατε, κύριε Πρόεδρε. Το Erasmus Plus είναι κάτι που το ζουν καθημερινά πάρα πολλοί πολίτες. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι συγγητής για συντάξει αυτής της νομοδότησης. Θέλουμε να φτάσει στο πλήρες δυναμικό του, το Erasmus Plus, και η Επιτροπή ΕΜΠΛ και Επιτροπικά ε, ε, ε, ασχολούνται με την έκθεση αυτή. Όπως γνωρίζετε, Μπορεί να μην συμφωνεί κανεί με τη μεθοδολογία, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως να επισημάνουμε τα ζητήματα που χρήζουν διορθώσεων, αλλά και να υπογραμμίσουμε ποιε είναι οι προτεραιότητές μα. Συναντηθήκαμε και με τους σκιώδεις συγκητές. Αρχή Σεπτεμβρίου ήρθε και η Κομισιόν και άλλοι ε, ενδιαφερόμενοι και πρέπει να πω ότι συμφωνήσαμε ότι είναι στη σωστή, στο σωστό δρόμο το Erasmus Plus, αλλά πολλά ακόμη μπορούν να βελτιωθούν. Τώρα, έρχομαι στη γνωμοδότησή μου. Έχω αναφέρει κάποιες προτεραιότητες αλλά είχα και πολύ περισσότερο αριθμό χαρακτήρων και τον ξεπέρασα, άρα πρέπει να τροποποιήσω ε, κάπως τη γνωμοδότηση. Η προτεραιότητά μας είναι η επαγγελματική κατάρτιση, θα πρέπει και στο Εράσμου να αντικατε... αντικατοπτρίζεται αυτό. Ε, πρέπει η, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση να αντικατοπτρίζει τις νέες ανάγκες. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνονται, πώς θα σχεδιάζεται η δακτέα ύλη και επίσης θέλουμε και ένα σύστημα μεταφοράς και αναγνώρισης μορίων. Επίσης ε, υπήρξαν κάποιες παραλήψεις που εντοπίσαμε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Erasmus ε, Plus. Θα πρέπει να δοθεί λοιπόν η απαραίτητη χρηματοδοτική υποστήριξη. Είναι πολύ σημαντικό, ιδίω σε πιο μικρούς δικαιούχους, σε άτομα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και όχι μόνο, ώστε ε, να μην μας διαφεύγει η πραγματικότητα και να μην υπάρχουν διακρίσεις. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόζονται ε, εναρμονισμένοι κανόνες με βάση ε, τα κοινά πρότυπα. Είναι σημαντικές ε, επίσης η, η απαραίτητη ενημέρωση για το job description, και η βελτιστοποίηση των ε, εργαλείων πληροφορικής, το εργαλείο κινητικότητα, το υπάλληλο. όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ώστε οι δικαιώχοι ε, να επωφεληθούν τα μάλα του προγράμματος. Και βέβαια θα πρέπει και η ανταλλαγή των πρακτικών να συνεχιστεί. Επίσης θα ήθελα να ε, υπάρξει ένα peer-to-peer review, ιδίως για τα θέματα κινητικότητας. Ευχαριστώ. Tom van den Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια και γενικότερα τους ε, εισηγητές που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, το Erasmus+. Ε, νομίζω ότι το δικό μας το καθήκον ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Erasmus Plus έχει ως στόχο να βελτιώσει τις δυνατότητες των νέων να βρουν θέση απασχόλησης. Εγώ προσωπικά ε, έχω ασχοληθεί με το Erasmus Plus, έχω σπουδάσει το πλαίσιο αυτού και γι' αυτό θέλω να κάνω κάποιες προτάσεις. Σήμερα το πρωί, παραδείγματος χάρη, επισκέφτηκα ένα πανεπιστήμιο το οποίο συμμετείχε στην επεξεργασία του νέου προγράμματος Erasmus+. Ε, κάτι που τους απασχόλησε πάρα πολύ ήταν ο έλεγχος της ποιότητας. Η ανταλλαγή φοιτητών θα πρέπει να έχει νόημα, ποιοτικά να είναι καλή και να είναι όλα τόσο καλά όσο και ε, στην πατρίδα του καθενός. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πούμε και στις ε, τροπολογίες. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να ε, αποκτώνται δεξιότητες και να πιστοποιούνται αυτές κατά τη διάρκεια του Erasmus Plus. Μετά ε, την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος πρέπει οι φοιτητές να μπορούν να βρουν θέση εργασίας. Χαίρομαι πάρα πολύ για την περαιτέρω συνεργασία. Και εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ Helga Stevens για το ισιά δεν είναι εδώ. Η Ρενάτε Βίμπα έχει το λόγο. Αλλά ούτε και αυτή είναι παρούσα. Γκονσάλες Πένας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ε, το στάκ της γνωμοδότησης ε, και για το έργο του και για την ε, επικοδομητική του προσέγγιση. Συμφωνούμε λοιπόν με την εστίαση, με το επίκεντρο της γνωμοδότησης και νομίζουμε ότι οι σημαντικές προκλήσεις είναι να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των ετούντων από τα διαφορετικά κράτη-μέλη, αφενός και αφετέρου οι ετούντες ε, θα πρέπει να έχουν επαρκή ενημέρωση για το πρόγραμμα. Βέβαια, υπάρχει και κάτι που μας ανησυχεί. Το πρόγραμμα Erasmus Plus να μην γίνει μεσοπρόθεσμα ένας δρόμος ε, που θα οδηγήσει ε, στην καθιέρωση, στην παγίωση ε, μιας επισφαλούς αγοράς εργασίας για τους νέους. Είναι δύσκολο αυτό. Αν δεν ενημερώνονται σωστά οι νέοι και για τα προγράμματα πανεπιστημιακής κινητικότητας, ούτε για τα προγράμματα επαγγελματική εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τις πρακτικές, όλα αυτά δημιουργούν επισφάλεια και ιδίως αν μιλάμε και για σπουδαστές με αναπηρία. 20.000 σπουδαστέ με αναπηρία. Ε, έχουμε στη χώρα μου. 13 μόνο πέρυσι είχαν πρόσβαση στο Erasmus Plus. Στο σχέδιο γνωμοδότηση γίνεται λόγο και για την εφαρμοστικότητα του προγράμματο. Είναι σημαντικό να μειώσουμε την ανεργία των νέων. Ναι, θα πρέπει όμω να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και στι πρακτικέ, ε, στα στάσει επιχειρήσει. Να μην γίνει αυτό τρόπο ε, αντικατάσταση εργαζομένων με επισφαλεί θέσει εργασία δηλαδή και καθόλου εγγύηση να προσλαμβάνονται για ένα συγκεκριμένο ε, διάστημα κάποιοι νέοι. Τον Νέγκρι είπε ότι πιο πολύ για την ένταξη των νέων θα πρέπει να νοηθεί το Erasmus Plus. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ένας χώρος ε, συναντήσεων, ε, σύμπηξη σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών λαών. Το Erasmus Plus πρέπει να το προωθήσουμε λοιπόν και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε για να μειωθούν οι ανισότητες και όχι το αντίθετο, να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες. Ευχαριστώ. Καρή δεν είναι εδώ. Η Λάουρα Τζέα δεν είναι εδώ. Τζο Εμελίν. Ντομινίκ Ματά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης για την έξι Πολιτισμού Ξέρουμε που εντάσσεται στην ενωσιακή αυτή προσέγγιση, μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών. Το ίδιο ισχύει για την εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτή η κινητικότητα θα έπρεπε να αφορά ε, όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, ώστε η κινητικότητα να μπορεί να προβλεφθεί στο μέλλον και οι άνεργοι να μπορούν να αναζητούν τελικά θέση εργασία σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες που έχουν έλλειμμα εργατικού δυναμικού. Επίσης βλέπουμε τα θέματα της επικαιρότητα ε, να παίρνουν μεγάλη διάσταση. Ε, επομένως, ο εισηγητής λέει ότι θα πρέπει και μιλάει για την ανάγκη οι μετανάστες να ενταχθούν. Όλος τυχαίως στο πρόγραμμα Erasmus Plus. Άρα το Erasmus Plus απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τον αρχικό του στόχο. Τέλος, εδώ πέρα ε, δεν αφήνουμε τίποτα. Επί παντός επιστητού ε, ασχολούμαστε. Δεν βλέπω να έχει δει κανείς άλλος το λόγο. Η Helga Stevens όμως ήρθε καθυστερημένα και έχει τώρα το λόγο για το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Βεβαίω, για κάθε θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να τη συγχαρώ για το πολύ καλό έγγραφο προσχέδιο. Είμαι πεπισμένη ότι με βάση αυτό το κείμενο μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και με τα χάρη συνεργαστώ μαζί της. Θα ήθελα να θέσω τα εξή σχόλια. Συμφωνώ απολύτως ότι το Erasmus Plus μπορεί να έχει θετική επίδραση στην απασχολησιμότητα. Έτσι, μας δίνει πολύ καλές δυνατότητες, μοναδικές δεξιότητες που μπορούμε να προσθέσουμε στην αγορά εργασίας. Όποιος ε, ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα μπορεί πιο εύκολα να βρει και δουλειά. Ε, οι αριθμοί δεν λένε ψέματα η επένδυση στο Erasmus Plus ε, αποτελεί επένδυση σε καλύτερους μισθούς. Βλέπω επίσης ότι από την έκθεση υπάρχει, ζητούμε μάλλον καλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και μεταξύ αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης. Συμφωνώ γιατί οι λάθος δεξιότητες έχει καταστροφικές επιπτώσεις για την αγορά εργασίας πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε και με αυτό το ζήτημα, ε, με τις ε, βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να εξάγει το καλύτερο αποτέλεσμα από κάθε μαθητή. Και έτσι να έχει και ο κάθε μαθητή τις ε, καλύτερε δυνατέ. ευκαιρίε. Θα ήθελα να κάνω και τι εξή προτάσει. Αυτή τη στιγμή το σημείο εστίαση στο Erasmus Plus αφορά περισσότερο ποσοτικούς στόχου. Όμως θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε την κατάλληλη έμφαση και στην ποιότητα. Δεν πρέπει να μιλούμε μόνο για τον αριθμό των ε, μαθητών ή φοιτητών που συμμετάσχουν στο Erasmus Plus. Και μετά για την προσβασιμότητα. Νομίζω ότι στην γνωμοδότηση πρέπει να ε, καλούμε για καλύτερη προσβασιμότητα στο πλαίσιο του Erasmus Plus. Αυτή τη στιγμή, ω προ την προσβασιμότητα, υπάρχουν ε, σημαντικά προβλήματα. Για παράδειγμα, ε, το δυσανάλογο διοικητικό άχθος ε, που πρέπει να επομίζονται άνθρωποι όπως εμένα για το κόστος των διερμηνέων τους, για παράδειγμα. Κλείνοντας, δεν μπορούμε να υποβιβάζουμε συγκεκριμένες ε, ομάδες πολιτών, λες και είναι λιγότερο σημαντικές. Πρέπει να γίνεται λόγος για άτομα με περιορισμούς και επαναλαμβάνω ότι είμαι διεθυμένη να συνεργαστώ για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. So, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καταληκτική ημερομηνία για την κατάσταση υπολογιών 29 Ανάτου το μεσημέρι. Θα αποφασίσουμε στις 8.11 στην Επιτροπή Απασχόληση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και τώρα ε, διάλειμμα. Το κερδίσαμε. Γιατί σας έχω πει ότι θα ξεκινήσουμε 5 παρατέταρτο. Οι καπνιστές θα με αποθεώσουν. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Ε, όσοι τους έκοψα το λόγο και τους είπα να βιαστούν, τους ζητάω συγγνώμη, ε, δεν μπορούσα και εγώ να το προβλέψω, λοιπόν μέχρι τις παρατέταρτο διάλειμμα.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

Dann starten wir in die Abstimmung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10. Πάμε στην ε, ψηφοφορία στο 10 EGF ε, εφαρμογές ε, καταρχήν ηλεκτρονικά για τη Microsoft από τη Φιλανδία παρακαλώ ψηφίσατε όλοι ως εκ τούτου έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίνεται. Πάμε στην περίπτωση EGF Ericsson από τη Σουηδία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πολύ ωραία. Σημείο υπαριθμών 11 Τη ημερήσια διάταξη νέε ευκαιρίε για τις μικρές επιχειρήσεις μεταφορών συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων. Ε, συμβαστική σε... αυτό τώρα... Κατά εγκρίνεται η συμβαστική εν υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική Δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην παράγραφο 1α νέο, τροπολογία 25, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, α, α, α νέα, η τροπολογία 8, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Ε, έκλεισε η ψηφορία. Εγκρίνεται. Η ου, η σημαστική ου, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική K K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4α αποσύρθηκε 4β, νιου, η 64 ε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, η 65 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, η 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η όμικρον, η συμβιβαστική, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 5 ανέα, 75, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η π, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η Q, υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Η R υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Η B υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Η Α, μισό λεπτό, η 7α νέα τροπολογία 89. Υπέρ παρακαλώ. Κατά ηλεκτρονική, ηλεκτρονική επαλήθευση. Η 89. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 90. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική. Α, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Μετά η τρία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα κατέπεσε, καταπίτη λέει ο πρόεδρος, εδάφιο ΑΑ. Η τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η οκτώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η εννέα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική τε ταφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 15 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά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 Dann ist aufgerufen die Nummer 12 in der Tagesordnung, European Semester for Economic Policy Coordination Implementation of 2006. Ευρωπαϊκό εξάμεινο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής εφαρμογής. Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική GA, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 19, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά πάμε στην τροπολογία υπαριθμών 25. Ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα της 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία υπαριθμών 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές ε, πρέπει να ε, Κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την τροπολογία υπαριθμών 28. Ψηφίσατε όλοι. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά αποχές, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 30 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 47. Ε, Σε δύο τμήματα, ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές, νομίζω απορρίφθηκε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Η 47, δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52. Πάλι Ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Για το πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά. Αχ, λέει ο πρόεδρος, πολύ δύσκολα σήμερα. Δεν βλέπω να παρακολουθήσω. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Άρα έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Εγκρίνεται. Η 54. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 54. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία 57. Υπέρ, κατά, αποχές. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 57. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. ή 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελικά δεν με πιστεύετε. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 58. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίφθηκε. Οι 59 και οι 60 είναι ίδιες υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η εν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 76 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 77 υπέρ, κατά, αποχές, ε, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, εγκρίνεται. Πάμε στο 79, υπέρ, κατά αποχές ε, ε, παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση για το 79 ψηφίσατε όλοι εγκρίθηκε στο 81 και 82 είναι ταυτόσιμες ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβαστική ή e, υπερκατά αποχές ε, γκρίνεται Πάμε στην 87, είναι μία προσθήκη στη συμβαστική 1, το δεύτερο τμήμα, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Μετά πάμε στην 93, ονομαστική ψηφορία, την έχουν ζητήσει οι σοσιαλδημοκράτες. Καταρχήν, ποιο συμφωνεί για αυτή τη διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας. Όποιος λοιπόν συμφωνεί πρέπει να σηκωθεί, να σηκωθεί όρθιος. είναι πάνω από ένα τέταρτο. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 93, πρώτο τμήμα, ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία, εγκρίθηκε. Πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, μου λένε. Ξαναψηφίζουμε για την 93 ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Για το πρώτο τμήμα, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τότε τώρα εγκρίθηκε κανονικά. Πάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα του 93 και εδώ πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, σηκωθήκατε όλοι πάλι πάρα πολύ καλά. Καλό αυτό για την υγεία. Κάτσε, σήκω, σήκω, κάτσε. Πάμε τώρα στην ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε την τροπολογία 95. Υπέρ. Κατά. Γιατί σηκώνετε τα χέρια σας. Ε, δεν νομίζω ότι είστε κουρασμένοι τέτοια ώρα. Ε, να σηκώνετε παρακαλώ τα χέρια. Ψηφίζουμε τώρα για την 95. Ψηφίζετε όλοι. Άρα τώρα ε, έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Πάμε στην 97. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και έχουμε τώρα ε, έτοιμα για ονομαστική ψηφοφορία από τους σοσιαλδημοκράτες για την 98 παρακαλώ. Πολύ ωραία. Ε, ψηφίζουμε λοιπόν για την 98. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε η ψηφορία. Εγκρίνεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 102. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 102. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 103 υπέρ, κατά, αποχές, η 104. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Επανεξετάζουμε την 104 επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Έκλειση ψηφορία. Υπέρ, κατά, αποχές για το δεύτερο τμήμα εγκρίθηκε. Η 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάσαμε στην 107 πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται. Εδώ για το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Νομίζω εγκρίθηκε Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές και αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε. Το τρίτο, ηλεκτρονική επαλήθευση ε, για το 107. Απορρίφθηκε. Η 108. 108 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε. 108 παρακαλώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμφωνήσατε όλοι. Πολύ ωραία. Η 109. Τροπολογία 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 110. Μισό λεπτό. 109. Ψηφίσατε όλοι. Η 110 υπέρ, η 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 112 ε, 112 πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. Υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Εκατόν δώδεκα. 112 παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Γιώτ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 118. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίθηκε. Η 119 υπέρ, κατά, ε, κατά. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Απορρίφθηκε. Πάμε στην 121. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Η L. Με προφορική τροπολογία. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 132. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η M συμβαστική υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίφθηκε ή 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 142 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πολύ ωραία. Απορρίφθηκε. 143 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 144. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 143. Ψηφίσατε όλοι, έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 144 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται ή 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα στα, ε, σε σκέψεις. Στην πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Στην τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, από ό,τι βλέπω ψηφίσατε όλοι. 35 ε, υπέρ, 12 κατά, 0 αποχές, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος των εργασιών μας, επόμενη συνεδρίαση 12 Οκτωβρίου και στις 13 ε, Οκτωβρίου το πρωί. Καλό βράδυ.